Funziona il microfono? Credo funzioni il microfono, c'era un po' di brusio, perciò non si... Eh, τα μικρόφωνα λειτουργούν παρά τις κάποιες παρεμβολές. Ξεκινάμε με το πρώτο σημείο λοιπόν στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ άλλων έχουμε και την έγκριση της ετήσιας έκθεσης για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών την έκθεση για τις δραστηριότητε του Ευρωπαίου Μεσολαβητή και τον ε, απολογισμό των δραστηριοτήτων του. Σήμερα έχουμε διερμηνία επίσης ε, σε όλες τις γλώσσες και web streaming και έχουμε πολλούς υπεύθυνους αναφορών από κάποιες από αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και επίσης να σας ειδοποιήσω ότι αύριο το πρωί στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης θα με αντικαταστήσει η συνάδελφος, ο αντιπρόεδρος κυρία Παλιαδέλη διότι πρέπει να παρευρεθώ σε μια διάσκεψη για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πρόεδρος της δικής μας Επιτροπής. Το σημείο 11 λοιπόν, οι ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών δεν θα συζητηθεί πρώτο, αλλά κατά τις 10 και 4. Το απόγευμα, όπως σας προειδοποίησα, θα μιλήσουμε και για την ε, έκθεση του κυρίου Μάγερ, την έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών, με αρκετές τροπολογίες, οι οποίες ήδη νομίζω κάποιες απλουστεύτηκαν, έχουν βρεθεί συμβαστικέ λύσεις και θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των τροπολογιών με κάποια σχόλια του εισηγητή πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα έχουμε επίσης και ανταλλαγή απόψεων για το έγγραφο εργασίας που έχει υποβάλει ο κ. Τουρκάης για την υλοποίηση τη οδηγία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε του υπεύθυνου των αναφορών που υπέβαλαν αναφορέ ε, στο σημείο 6, ε, 8 και 9 μαζί μα. Αύριο το πρωί, κατά τα άλλα, θα έχουμε τους αναφέροντες των σημείων 14, 15, 17, 18, 19, 20 και 21. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ωραία, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Έχει εγκριθεί λοιπόν. Σημείο δεύτερο, όπως σε κάθε συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής, έχουν μοιραστεί την περασμένη εβδομάδα μαζί με τις δικές μου ανακοινώσεις οι διαδικασίες λήξης αναφορών για τις οποίες δεν καταφέραμε να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες ε, για τους αναφέροντες, κάποιες οι οποίες έχουν παραμείνει εκκρεμείς ή σε τέλμα. Τέλος πάντων ε, υπάρχουν κάποιες αναφορές που διαθέτει στα χέρια της η γραμματεία. Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες για αυτές. Η στοιχεία θα έλεγα λοιπόν να εγκρίνεται και τις ε, προσαρτηθήσεις αυτές τις πληροφορίες. Δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις. Έχουν εγκριθεί και αυτές. Και εφόσον δεν έχω ανακοινώσει, περνάω κατευθείαν στο σημείο 4. Ξεκινάει η συζήτηση για την αναφορά 163 του 2010 που υπέβαλε Γερμανός υπηκό σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων. Ο αναφέρον δεν παρίσταται, οπότε θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον. Ε, με συγχωρείτε, η γραμματεία μου εξηγεί κάτι. Δεν θα συζητηθεί η αναφορά αυτή. Λάβαμε όμως για την αναφορά αυτή τη γνωμοδότηση, τη γνωμοδότηση της ε, νομικής υπηρεσίας, η οποία μοιράστηκε σε όλα τα μέλη, οπότε δεν θα γίνει τώρα συζήτηση. Απλώς προς ενημέρωσή σας, θα χρησιμοποιηθεί αυτή η πληροφορία για την αξιολόγηση της, της έκθεσης σε σχέση με την δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών. Για το σημείο λοιπόν αυτό, το πέμπτο, ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών, να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μέγερ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής για τις τροπολογίες που κατέθεσαν, τις 34 τροπολογίες τις οποίες αναφέρθηκε προηγουμένως η Πρόεδρός μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάν, τον κύριο Μποστινάρου, τον κύριο Σαλαβράκο, την κυρία Βέρτμαν, την κυρία Μπούλαντ και τη Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών γιατί όλες οι τροπολογίες αυτές ε, κατέβαλαν προσπάθεια να βελτιώσουν το κείμενό μου και προσπάθησα και εγώ να καταλήξω στη συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές σε μια σύμπνη για τα θέματα αυτά μέσα στα, στα πλαίσια αυτής της συνένεσης. Έχω συντάξει έξι συν... συμβιβαστικές ε, τροπολογίες που καλύπτουν πιστεύω το 90% των προτάσεων από τις διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες για συγκεκριμένα θέματα στα πλαίσια μιας προσπάθειας συμβιβασμού. Προφανώς η Επιτροπή μας είναι η πιο σημαντική και καταλληλότερη να, παρουσια... να παρακολουθεί τα θέματα των πολιτών. Θα πρέπει να του υποδεικνύει τρόπους για να αντιμετωπίσουν τις διεκδικήσεις των δικαιωμάτων τους και να υπάρχει μια ευρία γνώση μεταξύ των πολιτών για την ύπαρξη της Επιτροπής μας, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προωθήσει την ε, πρόσβαση στα έγγραφα. Θα πρέπει να υπάρξει και με συζήτηση για το θέμα της περιορισμένης σφαίρας εφαρμογής της Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επίσης είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί και η συνεργασία των κρατών μελών για το έργο της Επιτρόπης Αναφορών και να δοθεί και μεγαλύτερη διαφάνεια στην αντιμετώπιση των ε, αναφορών μέσω μιας απλοποίησης της εσωτερικής διαδικασίας στην Επιτροπή μας και μέσα στα πλαίσια μιας καλύτερης συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Όλες αυτές οι τροπολογίες έχουν γίνει δεκτές από τους βουλευτές που κατέθεσαν αντίστοιχες τροπολογίες, γι' αυτό θέλω δημόσια να τους αποτίσω φόρο τιμή και να του ευχαριστήσω γιατί αυτό απλοποίησε και έκανε πιο ε, εφικτή την εργασία μου και με τον τρόπο αυτό έχει εμπλουτιστεί το κείμενο χάρη στη συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων. Νομίζω ότι η συνένεση αυτή μπορεί σήμερα να υλοποιηθεί με την ψηφοφορία. Και τέλος θέλω να σας ανακοινώσω ότι παρουσίασε και μια προφορική τροπολογία στην εκθεσή μου, ώστε σε αιτιολογικές σκέψεις να περιλαμβάνεται και μια αναφορά στη γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής για την έκθεση 0163-2010 σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις προδικαστικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είναι ακριβώς το θέμα το οποίο μας απασχόλησε προηγουμένως. Αυτά λοιπόν και θα ήθελα κλείνοντα να ευχαριστήσω και πάλι όλε τι κοινοβουλευτικέ ομάδε για την συνένεση που έχουν επιφυλάξει σε σχέση με την εκθέσή μου. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία για την έκθεση του συναδέλφου Μέγερ. Τροπολογία 10 στην παράγραφο 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Παράγραφος 1α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 στην παράγραφο 1b. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 στην παράγραφο 1c. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τεχνική τροπολογία στην παράγραφο 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 στην παράγραφο 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 στην παράγραφο 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 στην παράγραφο 5α υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 στην παράγραφο 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 στην παράγραφο 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 στην παράγραφο 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 στην παράγραφο 10 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 23 και 24. 23 και 24 στην παράγραφο 11α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 25 στην παράγραφο 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 στην παράγραφο 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 στην παράγραφο 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 στην παράγραφο 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 στην παράγραφο 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 στην παράγραφο 25. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33. 33 υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε. Εκτός να επαναλάβουμε, υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται, εγκρίνεται 34 παράγραφος 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 τεολογικη σκεψη σκέψη 3α. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία εκ μέρους του εισηγητή. Αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Όχι. Δεν θέλει να την παρουσιάσει ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 για την αιτιολογική σκέψη α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. και άλλη προφορική τροπολογία από την ομάδα των φιλελευθέρων. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την παρουσίαση της προφορικής τροπολογίας. Θέλουν να την παρουσιάσουν οι εκπρόσωποι της ομάδας. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τροπολογία 4 όπως τροποποιήθηκε με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5, αιτιολογική σκέψη D, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία E, αιτιολογική σκέψη F, θα ψηφίσουμε κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επτά, για το νεοτιολογική σκέψη ΠΑ υπέρ. Κατά. Αποχές. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες για να ξαναψηφίσουμε. επτά λοιπόν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8. Αιτιολογική σκέψη S. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Αιτιολογική σκέψη T. Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στο συνάδελφο Μέγερ. Eh, και τώρα έχουμε τη συζήτηση υπό το σημείο 6, 273 του 2010, από την κυρία Μαρία Γκράτσια Κανούτη, αναφορά ε, για την οποία έχουν έρθει εδώ ο κύριος Πιετζόρτζο Τζόρτζο Μπενβενούτη, που εκπροσωπεί την Ένωση Οικολογικού Κινήματος της Αριλέγγιας Ιταλίας και του δίνω το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ για την προσοχή και τη δυνατότητα να συζητήσουμε εδώ, στην Επιτροπή αυτή, το δικαίωμα για ένα υγιές περιβάλλον. Το κίνημα της οικολογικής ε, Ιταλίας ασχολείται με το θέμα των χωματερών στην Ιταλία, ιδίως με το θέμα της Μαλαγκρότα κοντά στη Ρώμη. Εδώ έχουμε πολλές ε, αναβολές της πάυσης λειτουργίας της χωματερής, όμως υπάρχουν και σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και κίνδυνοι, επειδή ακριβώς προβλέπεται εκεί αυτός ο χώρος διάθεσης αποβλήτων και συγκεκριμένα σε ε, στο Λάτσιο, την ε, περιφέρεια αυτή, αυτές τις ημέρες συζητιέται για πολλωστή φορά το κατά πόσον θα δεν βρεθεί ένας αλλακτικός χώρος διάθεσης αποβλήτων ώστε να κλείσει τελικά η χωματερία αυτή. Κάθε Πολιτή έχει απαραβίαστο και αναφέρεται το δικαίωμα σε υγιέ περιβάλλον, όμω ε, στην περίπτωση των 350 περίπου χιλιάδων κατοίκων που βρίσκονται κοντά στη Μαρλαγκρότα, η αρχή αυτή παραβιάζεται συστηματικά. Γι' αυτό λοιπόν υποβάλαμε την αναφορά αυτή προ το Ευρωκοινοβούλιο, αναφορά για την οποία έχω έρθει σήμερα εδώ ώστε να προσπιστώ τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών ενώπιον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εγγυηθούμε την ε, προστασία των δικαιωμάτων για το υγιέ περιβάλλον. Δεν είναι καθόλου περιττό να θυμόμαστε ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα έχει αναλάβει εδώ σοβαρό ρόλο μέσω και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εγκρίνοντας τις αρχές της πρόληψης, της, ε, ε, του ρηπαίνοντος που πληρώνει και της ε, αποζημίωσης των βλαβών. Εδώ Υπάρχει και η οδηγία 4 για τους χώρους διάθεσης αποβλήτων του 1999 κάθετος 31 όπου υπάρχουν ε, υποσχέσεις και για μελλοντικού νόμους. Εκεί λέγεται ότι πρέπει να γίνεται διάθεση αποβλήτων με τρόπο ασφαλή και ελεγχόμενο. Είναι λοιπόν σημαντικό και σκόπιμο να ασχοληθούμε με την πρόληψη, την ανακύκλωση και την επαναξιοποίηση των αποβλήτων ώστε να εξοικονομήσουμε φυσικούς πόρους και να εξορθολογήσουμε τη χρήση της γης. Ε, ωστόσο δεν αρκεί αυτό, διότι ο κοινο... κοινοτικό νομοθέτης στην οδηγία 1999-31 έχει αναφερθεί και στις αρχές που εμπνέουν ε, την περιβαλλοντική μας δράση. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε εδώ με λεπτομερή τρόπο το όλο κείμενο, της τους κανόνες για να στυλιτεύσουμε τις ανεπάρκειες που έχουν διαπραχθεί στην περίπτωση της Μαλαγκρότα από τις σταλικές ε, Περιφερειακές Αρχές οι οποίες ε, θα πρέπει να δικαιολογήσουν τους σκοπούς που έχουν επιδιώξει υπό το πνεύμα αυτής της οδηγίας. Οι πολίτες που διαμένουν στην εν λόγω περιοχή εδώ και χρόνια συστηματικά ε, ζουν την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, την υγεία, του να ζουν σε ένα υγιές περιβάλλον. Η αναφορά που έχουμε ήδη υποβάλει αναφέρεται σε τρία συγκεκριμένα προβλήματα. Πρώτον, την ε, διάθεση μη επεξεργασμένων αποβλήτων ε, στον συγκεκριμένο χώρο, την απόρριψη ε, των αποβλήτων στον, στην περιοχή του ποταμού Γκαλέρια κοντά στην πρωτεύουσα, πάλι για ανεπεξέργαστα απόβλητα. Με συγχωρείτε, οι διερμηνείς δεν καταφέρουν να σας προλάβουν. Επίσης η παρουσία βουνών σκουπιδιών που βρίσκονται στην δημόσια οδό και δυσκολεύουν αναγκάζουν μάλλον σε παράκαμψη την ίδια την κυκλοφορία. Επίσης υπάρχει ένα πλαίσιο παρανομίας, το οποίο μόλις σας περιέγραψα και το οποίο επιδενώνεται έτσι περαιτέρω το γεγονός ότι οι Ιταλικές αρχές γνωρίζουν πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πλαίσιο το πλαίσιο που δημιουργείται από το χώρο διάθεσης της Μαλαγκρότα για τους πολίτες που διαμένουν σε αυτή την περιοχή. Παρ' όλα αυτά παραμένουν ε, αδρανείς. Ο Οργανισμός για την Προστασία του Περιβάλλοντος, η Παλάτσιο, έχει ήδη πιστοποιήσει σε πρόσφατη μελέτη ότι υπάρχει ρήπανση των υδροφόρων οριζόντων και των υδάτων της επιφάνειας στην περιοχή του χώρου διάθεσης της Μαλαγκρότα. Εκεί φτάνουν διάφορες ε, υδάτιν, διάφοροι υδάτινοι δρόμοι, ε, περιφερειακοί, οι οποίοι καταλήγουν όμως να ρηπαίνουν και τη Ρώμη. Και επίσης ε, με το Προεδρικό Διάταγμα 334 της 16ης Αυγούστου του 1999, ε, ταξινομήθηκε η περιοχή της Μαλαγκρότα ως επικίνδυνη περιοχή ε, από περιβαλλοντική άποψη που μπορεί να δημιουργήσει και περιβαλλοντικέ κρίσει. Η ίδια Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση με διαδικασία επί για παραβίαση τη συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση εκατά ε, της Ιταλίας, η οποία όμως εκμοδίκησε από το 2008 επειδή είχε υποβληθεί ένα σχέδιο προσαρμογής ε, της χωματερής, το οποίο όμως για την ώρα έχει μείνει στα χαρτιά, είχε ε, αντιληφθεί την έκταση του προβλήματος, του προβλήματος που θέτει ο χώρος διάθεσης της Μαρλαγκρότα. Τα συμπεράσματα τώρα. Για όλους τους νομικούς λόγους που προανέφερα και επειδή ισχύει η, το απαραβίαστο του δικαιώματος ε, στο υγιές περιβάλλον των πληθυσμών που κατοικούν στην περιοχή της Μαλαγκρότα, και επειδή δεν προβλέπεται η άμεση προσαρμογή του χώρου διάθεσης της Μαλαγκρότα και την ε, το ενάμεση πάυση λειτουργία της χωματερή αυτής και την ε, βελτιστοποίηση της περιοχής της Μαλαγκρότα, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, ε, ήδη είχε δοθεί υπόσχεση γι' αυτό τον Απρίλιο του 2011 και επειδή δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις που να επιτρέπουν τη λύση του προβλήματος της Μαλαγκρότα. Απευθύνω την έκκληση των πολιτών μας και της Ένωσης Ιτάλια Σολιντάλια, της Αλληλέγγυας Ιταλίας προς την κοινότητα, ώστε εμπνεόμενοι από όλες τις αρχές για την περιβαλλοντική δράση να ε, παροτρύνουν ή να επιβάλλουν στις Ιταλικές αρχές να εγκρίνουν τα απαραίτητα μέτρα. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών, χωρίς να αναβληθεί ξανά η παρέμβαση που σήμερα δεν μπορεί πλέον να αναβληθεί. Είναι απαραίτητη. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ενημερώνω ότι η Επιτροπή για τη σημερινή συνεδρίαση, η Γραμματεία μάλλον της Επιτροπής, έχει προσκαλέσει εκπροσώπους ε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των δημοτικών αρχών, των περιφερειακών αρχών της Ρώμης και εκπρόσωποι των ε, έχουν έρθει εδώ κάποια μέλη των αρχών αυτών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον Κλάουντιο Βεσέλη, ο οποίος εκπροσωπεί την ε, περιοχή της Ρώμης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, εκπροσωπώ τον ε, νομάρχη της περιοχής της Ρώμης. Ασχολούμαι με τα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας σε αυτή την περιοχή και σε ό,τι αφορά το χώρο διάθεσης της ε, Μαϊλαγκρότα, μια από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης όπου προβλέπεται μια μελλοντική προέκτασή της τουλάχιστον σε 200 εκτάρια. Στα δυτικά λοιπόν της Ρώμης, στην περιοχή του Λάτσιο, εδώ χρησιμοποιείται ο χώρος αυτός για διάθεση ανεπεξέργαση των αποβλήτων που προέρχονται από την πρωτεύουσα, την πόλη του Βατικανού και των γειτονικών πόλεων ε, όπως το Φιωμιτσίνο. Εδώ μιλάμε για μια λεκάνη όπου κατοικούν τουλάχιστον 300.000 πολίτες. Η διαδικασία της διάθεσης των αποβλήτων που ξεκίνησε το 1995 στην χωματερή αυτή ε, αναβλήθηκε, συνεχίστηκε μάλλον μέχρι να εντοπιστεί ένας εναλλακτικό χώρος διάθεσης, επεξεργασίας των αποβλήτων επίσης, τα οποία ε, προκύπτουν από το προεδρικό διάταγμα του νομάρχη της περιοχής του Λάτσιο, από τον Σεπτέμβριο του 2010. Για την ώρα ακόμη ε, κινείται η διαδικασία ώστε να προκύψει από τις αρχές του Λάτσιο η έγκριση για να βρεθεί ο εναλλακτικό χώρος διάθεσης. Στις 4 Μαΐου του περασμένου του 2011 συζητήθηκε τελευταία φορά το θέμα αυτό και πέραν των ε, κοινοτικών, τομεακών και εθνικών μας νόμων ε, προβλήθηκαν ε, τα εξή επιχειρήματα. Με το διάταγμα 26 του 1995 και όπως προβλέπει το κοινοβουλευτικό ο νόμος 36 του 2003 για την υλοποίηση της οδηγίας 31 του 1991 προκειμένου να μην υπάρχει περιβαλλοντική ρήπανση ή βλάβη για την ανθρώπινη υγεία πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Ο, το είπε όμως αυτό και πρόσωπος της Ένωσης που προηγήθηκε. Το σχέδιο αυτό πάυσης λειτουργίας, η προσαρμογή στις χωματερίες παρέμεινε νεκρό γράμμα. Ε, στη δεκαετία του 90 η διάθεση των αποβλήτων και το πρόγραμμα αυτό έγινε μέσω ενός προγράμματος που ονομάστηκε Polder, με ένα τσιμεντένιο τοίχο που περιέφρασε την ε, χωματερή ώστε να προστατεύεται και το αργυλώδες χώμα της, ε, του εδάφους. Αυτό όμως ε, πέραν του διαφράγματος εντός και εκτός του χρησιμοποιήθηκαν και επιπλέον ζώνες ώστε να μπορούν να γίνουν μετρήσεις του υδροφόρους ορίζοντες, και αναλύσεις στο νερό για βακτηριολογικές και μικροβιολογικές αναλύσεις. Η χωματερή, όπως προβλέπει ο νόμος, διαθέτει ένα σύστημα κατακράτησης των βιοαερίων που προέρχονται από την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και σύστημα παραγωγής μεθανίου μέσω της χρήσης των αποβλήτων. όλα αυτά όπως ορίζει ο νόμος για το θέμα αυτό. Το θέμα της χωματερής στην ε, νομοθεσία 46 του 2003 απαιτεί και διαδικασίες επιθεώρησης και ελέγχου. Όλα τα μέτρα λοιπόν πρέπει να προβλεφθούν ώστε να μην υπάρξουν ατυχήματα λόγω της λειτουργίας του χώρου διάθεσης και να προστατευτεί το περιβάλλον από ενδεχόμενους κινδύνους ε, ρήπανσης. Ε, σημασία έχει και η συστηματικότητα των ε, ελέγχων Υπάρχουν δύο κεντρικοί σταθμοί για την παρακολούθηση της περιοχής, τις κλιματολογικές ε, συνθήκες, ενώ η ποιότητα των υπογείων υδάτων ελέγχεται με τις ε, συστηματικές αναλύσεις που γίνονται είτε από τον διαχειριστή της χωματερής είτε από τις περιφερειακές αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος, με δείγματα τα οποία ε, λαμβάνονται υπογείως. η υπέρβαση των επιτρεπτόμενων όριων για το νικέλιο, το σίδηρο, τον υδράργυρο ε, έχουν ήδη διαπιστωθεί, ενώ η εταιρεία Τζόβι που είναι υπεύθυνη για την διαχείριση της χωματερής ασχολήθηκε και με άλλες ε, πηγές ε, που διαθέτουν τα προβλήματά τους στο χώρο αυτό. Η αρχές της περιφέρειας του, της, του νομού του Λάτσιο έλαβαν γνώση για την υπέρβαση των ορίων αυτών και πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία για το ποιες είναι οι πηγές της ρήπανσης αυτής. Η περιοχή όπου εντοπίζεται η εν λόγω χωματερή μοιράζεται το χώρο αυτό με άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως τα δηληστήρια πετρελαίου, τις χώρους επεξεργασίας των αποβλήτων, εξορρυκτικές δραστηριότητες, γεωργικές, ε, κτηνοτροφικές και δρόμους ε, κυκλοφορίας οχημάτων, στοιχεία που όλα αυτά μπορούν να επιβαρύνουν ε, το περιβάλλον. Το Ανώτατο Ίδρυμα για την Έρευνα και την Προστασία του Περιβάλλοντος ερεύνησε την περιοχή της Μαλαγκρότα και το Υπουργείο του Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε με προηγούμενους ελέγχους ότι υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικός σε ολόκληρη την περιοχή. Συγκεκριμένα λόγω της ποιότητας των ε, υδάτων επιφανείας και των υπογείων υδάτων. Τα δείγματα ε, των ατμοσφαιρικών αερίων όμως και η μελέτη των νερών έδειξαν ότι ακόμη και η κυκλοφορία οχημάτων ή η βιομηχανική μόλυνση επιβαρύνουν την κατάσταση. Η μελέτη που διεξήχθηκε λόγω τη μεγάλη έκταση τη περιοχής που ερευνήθηκε, αλλά και τη πολυπλοκότητα των όλων πηγών της ρήπανση, που μπορεί να έχουν συνδυαστεί και μεταξύ τους δεν επέτρεψε να πιστοποιήσουμε αν η ρήπανση την οποία συζητούμε οφείλεται στο διάθεση των αποβλήτων σε αυτή την περιοχή. Πάντως, ως σήμερα, είτε με βάση τις ε, διεξαχθήσεις μελέτες από τα όργανα ελέγχου, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε την ε, σχέση αιτίας-αιτιατού μεταξύ της ρήπανσης και του χώρου διάθεσης με το ευρύτερο περιβάλλον στην όλη περιοχή. Πάντως, <clears throat> υπάρχουν και καύσιμα στα υπόγεια ε, ύδατα, δείγματα καυσίμου στα υπόγεια ύδατα, που δείχνουν ότι από τα πηγάδια της περιοχής μπορεί να έχει προέλθει μόλυνση, που δεν σχετίζεται αναγκαστικά άμεσα με το χώρο διάθεσης της Μαλαγκρότα. Πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον ε, είναι αξιόπιστα τα δείγματα των ε, περιβαλλοντικών αναλύσεων. Πρέπει να υπάρξει σαφής διασύνδεση των αιτίου αιτιατού μεταξύ των υδροφο... της, της ρήπανσης των ε, υδροφόρων οριζόντων και της δράσης της, χωμα... της λειτουργίας της χωματερής από τον Σεπτέμβριο του 2010 με το διάταγμα 255 ο Δήμαρχος της Ρώμης ε, ζήτησε την μελέτη για τη, λήψη επιγόντων, τη μελέτη της λειτουργίας της κομματερής αυτής και τη λήψη επιγόντων μέτρων. Κλείνω λέγοντας ότι για να έχουμε ένα πλαίσιο νομικής ε, βεβαιότητας και ρυθμιστικής βεβαιότητας σε σχέση με τη ρήπανση της ε, ευρύτερης περιοχής Ήδη τις τελευταίες μέρες η Περιφέρεια Λάτσιο, η Κοινοτική Αρχή της Ρώμης και ο Δήμαρχος της Ρώμης υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεννόησης για την πραγματοποίηση έρευνα στην περιοχή της Μαλαγκρότα ώστε να διατεθεί ένα κονδύλι 3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και με την ελπίδα ότι με τη συνεργασία των δημοτικών οργάνων ελέγχου και των εθνικών θεσμικών οργάνων, όπως η ΙΣΠΡΑ, το Οργανισμό για την Προστασία Περιβάλλοντος, το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών, με, όλη, με τη συνεργασία όλων αυτών των φορέων, να μπορέσουμε να δώσουμε μια βέβαιη απάντηση για το ποιοι είναι, ποιες είναι οι πραγματικές πηγές της ρήπανσης και να βρεθούν πραγματικοί αυτούργοι. Ρήπανση η οποία αναμφισβήτητα υπάρχει στην περιοχή της Μαλαγκρότα. Αλλά έως σήμερα δυστυχώς δεν μπορεί να διασυνδεθεί με απόλυτη νομική όχι τόσο επιστημονική, αλλά νομική βεβαιότητα με την ε, λειτουργία της ε, χωματερής. Διότι ως τόσο η δικαστική λειτουργεί όσο και οι ελεγκτές αυτή τη στιγμή κάνουν ό,τι μπορούν για να αναλάβουν πλήρω τι ευθύνε του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Μαγκανάρο για να ακούσουμε περισσότερο για την έρευνα που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα το 2009. Σε σχέση με την, ε, το χώρο απόρριψης της Μαλαγκρότα, και το 2010 έρθει σε επαφή με τις Ιταλικές αρχές, οι οποίες συνεχίστηκαν και το 2011. Η τελευταία φορά που αναφέρθηκε από την Επιτροπή, το θέμα στην Επιτροπή Αναφορών τον Ιανουάριο του 2011 για τη Μαλαγκρότα, ήρθαμε και πάλι σε επαφή με τις Ιταλικές αρχές, οι οποίες μας έστειλαν διευκρινιστικές πληροφορίες στο τέλος του 2011 και στη, του Ιανουαρίου 2011 και το Μάρτιο. Βέβαια δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που είναι ακόμα εν εξελίξη. Είναι πολύ πιθανό ότι η Κομισιόν θα πρέπει να, η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να καταλήξει σε μία απόφαση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, κάποιοι οποίοι θα θέλανε να λάβουν το λόγο μεταξύ των κοινοβουλευτικών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά μου φαίνεται ότι θα πρέπει να το ακούσουμε και κάνω μια έκκληση, με κάνω μια παράκληση προς την Επιτροπή. Οι επικρίσεις, οι αναφέροντες ε, έχουν αναφέρει διάφορα σημεία θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, να δούμε δηλαδή ποια είναι τα αποτελέσματα που ενδεχομένω μπορεί να μας υποβάλει η Επιτροπή. Προς το παρόν πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση αρκετά ε, σοβαρή και ελπίζω και ζητώ από την Επιτροπή να πάρει πολύ σοβαρά υπόψη αυτά που αναφέρουν οι ε, υποβάλλοντες στην αναφορά. Uh, uh, uh, Ήταν πολύ καλή αυτή η πρόταση, την οποία θέλω και εγώ να υποστηρίξω. Εντάξει. Κυρία Άικεν, και εγώ συμφωνώ. Απλώς, η εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι αμφισβητείτε το ότι υπάρχουν προβλήματα με τον χώρο απόρριψης, με τη χωματερή, αλλά Ακόμα και αν πείτε ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες πηγές ρήπανσης, φανταζούμε ότι δεν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη χωματέρη. Δεν πρέπει να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου θα πούμε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε όλες τις πηγές της ρήπανση, να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όλα δεν είναι καλά με το χώρο απόρριψης της Μαλαγκρότα. Ελπίζω ότι δεν θα καταλήξουμε στο σημείο αυτό, γιατί αυτά τα οποία είπαν οι αρμόδιες Ιταλικές Αρχές ήταν λιγάκι ασαφείς για το θέμα αυτό. Άλλες παρεμβάσεις. Η κυρία Μέρκης και πάλι. Για τον αναφερόμενο θα ήθελα να πω ότι έχουμε λάβει πολλές αναφορές από την Ιταλία, πολλές φορές που αφορούν, πάρα πολλές από τις οποίες αφορούν το ίδιο αυτό θέμα. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι πράγματι θέλουμε να προχωρήσουμε σε βάθος και να κατανοήσουμε πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα και στη συνέχεια να το φέρουμε στο προσκήνιο και να, <clears throat> να συνεχίσουμε τη συζήτηση σε ένα συνολικό επίπεδο. Επομένως, θέλω να τονίσω ότι ο στόχος μας δεν είναι να ξεπετάξουμε μέσα εισαγωγικά αυτή την αναφορά. Αντίθετα, θέλουμε να δώσουμε την πρέπει προσοχή στο πρόβλημα αυτό και από αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής με την γενική πολιτική ε, για τις ε, χωματερές και τις απορρίψεις θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Θέλουν οι υπογράφοντες την αναφορά να επανέλθουν. Θέλετε να απαντήσετε για καταρχήν ο εκπρόσωπος της επαρχίας να λάβει το, το λόγο. Θα ήθελα να σας πω ότι λυπάμαι αν δόθηκε η εντύπωση ότι υπήρχε κάποια διστακτικότητα από την πλευρά των επαρχιακών αρχών. Εμείς έχουμε απόλυτη επίγνωση των προβλημάτων που συνάπτονται με την χωματερία αυτή, αλλά για να μπορέσουμε να δράσουμε κατά του διαχειριστή του χώρου αυτού απόρριψης θα πρέπει να έχουμε αδιάσυστες, ε, αδιάσυστα στοιχεία, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι το έχουμε. Επομένω, δεν μπορούμε, επί τη βάση των στοιχείων που έχουμε για την ρήπανση, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια σαφή αιτιακή σχέση μεταξύ της, ε, ε της χωματερής και της ρήπανσης. Και το αρμόδιο δικαστήριο είπε ότι θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει σαφής ευθύνη του διαχειριστή της, ε, του χώρου απόρριψης αν είναι να προχωρήσουμε στη λήψη κάποιων μέτρων. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα με τα αστικά απόβλητα τα οποία υπάρχουν συσσωρευμένα εκεί. Δεν είναι λαθασμένο να πούμε ότι έχουμε ενώπιόν μας ένα τέρας ουσιαστικά, μία ε, συσσόρευση αποβλήτων από 3 εκατομμύρια κατοίκων. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι παρά την ευρωπαϊκή οδηγία και τις ε, ευρωπαϊκές και τις ιταλικές οδηγίες που εφαρμόσουν την ε, Ευρωπαϊκή Οδηγία έχουμε ακόμα δυστυχώς στην ε, Ρώμη μία συλλήβδην συλλογή στοιχείων απορριμμάτων. Ένα πολύ μεγάλο μέρος λοιπόν των ε, απορριμμάτων δεν τυχάνουν ανακύκλωση ή επιλεκτική συλλογή, αλλά καταλήγουν όλα σε αυτή τη χωματερία. Αυτό φυσικά σημαίνει σημαντικά προβλήματα για τους ε, κατοίκους της περιοχής της, ε, του χώρου απόρριψης και αυτή τη στιγμή εφόσον δεν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια σαφής παραβίαση της οδηγίας δεν μπορούμε να προχωράσουμε περισσότερο αλλά θα μπορούσε με μια καλύτερη επιλεκτική συλλογή των αποβλήτων να προχωρήσουμε στο κλείσιμο αυτής της ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, όπως προσπαθήσαμε να δείξουμε, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο κρατάει εδώ και δεκαετίε, δεν είναι σημερινό. Από το πρόβλημα αυτό, για το πρόβλημα αυτό λοιπόν νομίζουμε ότι οι δημοτικές αρχές της Ιταλίας και οι περιφερειακές αρχές θα έπρεπε να έχουν βρει λύση εδώ και 10 χρόνια. Τώρα, κατά τα άλλα, οι ευθύνε. Ε, μάλλον το πρόβλημα δεν είναι να γίνει πύριψη ευθυνών εδώ με μια δειγματοληψία το κατά πόσον υπάρχουν άμεσες ευθύνες ή όχι είναι κάτι που μπορεί να λυθεί στην Ιταλία. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτή την περιοχή η οποία είναι τεράστια σε έκταση και με εγκαταστάσεις που όλες έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο πολύ σημαντικό και με πολύ διαφορετικές δραστηριότητες, διαφορετικών κατηγοριών. Είναι λοιπόν αδύνατο να κλείνει κανείς τα μάτια και να λέει ας φτιάξουμε κι άλλη μία χωματερή στην ίδια περιοχή με αυτό το χώρο διάθεσης αποβλήτων. Όπως έλεγε και ο εκπρόσωπος της περιφερειακής μας αρχής, της επαρχίας μας, ε, η Ιταλία θα πρέπει να προσαρμοστεί και με το είδος των χώρων διάθεσης που έχουν πλέον ξεπεραστεί. Ε, θα πρέπει να δούμε και το πρότυπο του Σαν Φραντίσκο. Δηλαδή να διακρίνουμε μεταξύ αποβλήτων ε, και να φτάσουμε και σε μηδενική επιβάρυνση από απόβλητα, ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία των συμπολιτών μας σε μια τόσο ευρεία περιοχή όπως αυτή της Μαλαγκρότα. Σας ε, ευχαριστώ. Ήθελε και ο συνάδελφος, η συνάδελφος το λόγο. Πολύ σύντομα προς τις αρχές, τους υπεύθυνου των αρχών. Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι παράνομο, λέτε, αλλά πιστεύετε ότι για την Ευρωπαϊκή Οδηγία των αποβλήτων βρίσκεστε στο ύψος των προσδοκιών, διότι εξ όσων ακούω, καθόλου δεν εκπληρώνονται οι απαιτήσει της οδηγίας. Γι' αυτό και στρεφόμενοι προ την Επιτροπή λέω ότι και η Επιτροπή θα έπρεπε να λάβει γνώση. Δεν είναι ένα θέμα ούτε εκλογικό ούτε ιδιωτικό για να αποφασιστεί εδώ τι είναι νόμιμο και τι όχι. Είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι σαφώ λοιπόν στην απάντησή σα, δεν είναι σαφέ, ε, εάν το βλέπετε το πρόβλημα ω ε, μια τοπική ιστορία. Λέτε έχουμε κάποιους νόμους που εδώ και πολύ καιρό δεν έχουν ε, εφαρμοστεί σωστά και οι έλεγχοι, πρέπει να κάνουμε σωστούς ελέγχους και τι θα συνεχίσετε. Όλοι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και νομίζω ότι μου θυμίζει πάρα πολύ όλα αυτά όσο έχουν γίνει στην καμπανία. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο, κύριο συνάδελφο Θέλω να προσθέσω κάτι. Είμαι σίγουρος ότι όταν μας προσθέσουν τα στοιχεία που λείπουν η Επιτροπή θα στηρίζονται και θα βασιστούν στη σαφή επιστημονική ανάλυση που πρέπει να γίνει. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, έλλειψη διαφάνεια αυτή τη στιγμή. καθότι βλέπουμε ότι από τη μια μεριά αυτοί που πιστεύουν ότι δηλητηριάζουν τα απόβλητα, τα ύδατα και η άλλη πλευρά που θεωρεί ότι δεν δηλητριάζονται, ότι δεν ρηπαίνουν, αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί αν δεν γίνει μια συγκεκριμένη ανάλυση της ποιότητας των υδάτων. Εγώ θέλω να ξέρω, υπάρχει ή δεν υπάρχει κάτι που ρηπαίνει. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε εάν δεν υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη έρευνα και αυτό βάσει επιστημονικών στοιχείων. Από τη στιγμή που υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλημα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι και είναι πολύ συγκεκριμένα τα βήματα. Το πρώτο βήμα είναι μια ανάλυση. Χωρίς το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης δεν μπορούμε να αποφαθούμε. Προς το παρόν υπάρχουν ε, κάποιες υπόνοιες, ε, κάποιες ε, κατηγορίες, αλλά επειδή πρόκειται για θέματα που πλήττουν την υγεία των κατοίκων, είναι πολύ σημαντικό να αποφανθούμε. Περασματικά δεν έχει εξαντληθεί το θέμα της αναφοράς. Θα έχουμε ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε, δεδομένης και της απάντησεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που μετά τις παρεμβάσεις που ακούσαμε θα ζητήσουμε να μας δώσει και κάποια παλιτέρω στοιχεία. Πρώτα απ' όλα απαντήσεις για το ότι αφορά, με τη, συμμόρ... ότι αφορά τη συμμόρφωση, για τα ειδικά μέτρα των ευρωπαϊκών οδηγιών, των σχετικών οδηγιών και για το περιβάλλον και για τα απόβλητα. Έπειτα την ανάγκη να γίνει αναλυτική επαλήθευση, επιστημονική επαλήθευση όλων των στοιχείων και θα προσθέσω εδώ και μια δική μου παρατήρηση ότι η παρέμβαση αυτή, η επιστημονική επαλήθευση από την πλευρά της Επιτροπής θα πρέπει να λάβει υπόψη και να μας ενημερώσει για τόσα συμβαίνουν και μετά από όσα μας είπε ο υπεύθυνο της Αρμοδίας Επιτροπής από την ε, Περιφερειακή Αρχή. Δηλαδή διαχείριση των αποβλήτων κατά τρόπο που να διατίθενται έτσι ώστε να δημιουργούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα ε, που ανέφερε και η Επιτροπή. Δηλαδή, ο πλήρης κύκλος διαχείρισης των αποβλήτων και ο σεβασμός ε, των ε, κανόνων των ευρωπαϊκών οδηγιών και αυτά που προβλέπουν σε σχέση με τη μείωση των αποβλήτων και όλα τα υπόλοιπα. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να τα λάβει όλα αυτά υπόψη όταν μας δώσει μια απάντηση. Ελπίζουμε αρκετά σύντομα ώστε να έχουμε και για αυτά διευκρινήσεις. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λοιπόν θα έλεγα να κλείσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ τους αναφερομένους και τους εκπροσώπους των αρχών της ωραίας επαρχίας της Ρώμης για την παρουσία τους. Θα σας τηρούμε ενήμερους για τις περαιτέρω εξελίξεις. Σημείο 7. Έκθεση σε σχέση με την εφαρμογή τη οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων. Παρόμοιο θέμα. Βάσει των αναφορών που ελήφθησαν εισηγητή ο συνάδελφο Τουργκάη, ο οποίο θα μα παρουσιάσει το εν λόγω έγγραφο. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι σαν εισηγητής για τα θύματα διαχείρισης των αποβλήτων θέλω να σας παρουσιάσω το έγγραφο εργασίας το οποίο έχει, έχω εκπονήσει σε σχέση με την οδηγία της διαχείρισης των αποβλήτων. Το έγγραφο αυτό έχετε ήδη στα χέρια σας ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη μητρική σας γλώσσα. Θα ήθελα να παρουσιάσω τα προκατακτικά συμπεράσματα που χαρακτηρίζουν το πρώτο στάδιο της εργασίας μας. Η πρόθεσή μου τόσο για σήμερα όσο και για αύριο ε, θα ήταν να υπάρξει μια ανοιχτή συζήτηση σε σχέση με την γραμμή εργασίας και γραμμή πλεύσεως που χρησιμοποίησα στην έκθεση αυτή και τις βασικές αρχές που διέπουν την έκθεση αυτή. Και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας και ποια σημεία θεωρείτε ότι πρέπει να είναι τα πιο προεξάρχοντα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να παρουσιάσουμε σε κάθε συζήτηση και σε συνάρτηση με την έκθεση που έχει γίνει η θεματική ομάδα μελέτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα θέματα διαχείρισης των αποβλήτων και που θα δημοσιευτεί πιστεύω πριν από την επόμενη συνεδρίασή μας τον Ιούλιο για να καθορίσουμε και τη γραμμή μας σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων. Ο στόχος μου λοιπόν είναι να εξασφαλίσω ότι θα υπάρξει εμπλουτισμός του γράφου εργασία σε σχέση με τρία θέματα. Πρώτον, επί τη βάση των συμπερασμάτων στα οποία θα καταλήξουμε σε αυτή τη συζήτηση. Δεύτερον, από αυτά τα οποία θα προκύψουν μετά τη συνάντησή μου αύριο με τους κοιόδης εισηγητές. Και τρίτον, επί τη βάση των συμπερασμάτων και των πορισμάτων της μελέτης, της ε, εξωτερικής μελέτης που θα γίνει υπό την αιγίδα της θεματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει όλων αυτών λοιπόν θα γίνει η συγγραφή του πρώτου σχεδίου εκθέσεως για να παρουσιαστεί ενώπιον όλων των συναδέλφων τον Οκτώβριο. Ελπίζω ότι αυτή η διαδικασία σας ικανοποιεί και γι' αυτό θα ήθελα να σας δώσω τις προκατακτικές, τα προκατακτικά μάλλον συμπεράσματα του εγγράφου εργασίας. Αυτά τα προκατακτικά συμπεράσματα ξεκινούν από το γεγονός ότι όλοι έχουμε αναγνωρίσει ότι οι περισσότερες αναφορές που έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορούν θέματα του περιβάλλοντο και μέσα στις αναφορές αυτές του περιβάλλοντος τα θέματα διαχείρισης των αποβλήτων είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπό μας. Από την έναρξη ήδη της έκτης κοινοβουλευτικής περίοδου του Κοινοβουλίου το 2004 ως το τέλος του 2010 η Επιτροπή μας εξέτασε 114 αναφορές σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. Σε μεγάλο βαθμό ο υψηλός αυτός αριθμός αναφορών καταδεικνύει χωρίς καμία αμφιβολία το γεγονός ότι τα απόβλητα δημιουργούν πολλές ανησυχίες στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά τονίζει και τη σημασία που έχει το θέμα αυτό στην καθημερινή του ζωή. Από την άποψη της Ευρωπαϊκής, από την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση της ποσότητας αποβλήτων. Ιδίω σε σχέση με τα απόβλητα τα οποία δεν είναι ανακυκλώσιμα ή αναχρησιμοποιήσιμα. Ο στόχος λοιπόν είναι να αναστραφεί η ιεραρχία των αποβλήτων. Αντί να μιλάμε για την απόρριψη των αποβλήτων, να μιλάμε για την πρόληψη των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίησή τους, την ανακύκλωσή τους ή ακόμα και την παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα. Αυτή λοιπόν είναι και η άποψη που περιλαμβάνεται στην Οδηγία 2008-98 της Ευρωπαϊκής Ένωσης τούτου λεχθέντος τώρα. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε. Πρώτα απ' όλα ότι τα κράτη-μέλη είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στον τομέα των αποβλήτων. Δεύτερον, ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει χρηματοδότηση για τη βελτίωση της υποδομής διαχείρισης των αποβλήτων. <clears throat> και, το... και αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να έρχεται από το Ταμείο Συνοχής ή από το... την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τρίτον, τα σχέδια τα οποία είναι πιο κατάλληλα για κοινοτική χρηματοδότηση θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ε, ρήτρε της οδηγίας. Τέταρτον, η μη εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιου για τα απόβλητα από την πλευρά των κρατών μελών είναι μια μεγάλη πρόκληση για την εφαρμογή των κοινοτικών αρχών που έχουν να κάνουν με τα απόβλητα. Πέμπτον, θα πρέπει η Επιτροπή να έχει περισσότερους πόρους για καλύτερη εποπτεία και αστυνόμευση των πολιτικών στον τομέα των αποβλήτων. <clears throat> Έκτον, πρέπει να βελτιώσουμε το διάλογο με του εμπλεκόμενου πληθυσμού και θα πρέπει οι πολίτε να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίε και του μηχανισμού διοικητικού και δικαστικού ελέγχου. Εβδόμο, θα πρέπει να προωθήσουμε μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και τη Επιτροπή Αναφορών, τη δική μα Επιτροπή, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη υπηρεσία που παρέχουμε στους πολίτες, καλύτερες απαντήσεις που δίνουμε στους αναφερόμενους και εν γέννη στους πολίτες. Αυτά λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι και κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι μπορούν να είναι οι οδηγές γραμμές, οι κύριοι πυλώνες επί των οποίων θα βασιστεί η έκθεση <clears throat> την οποία εγώ θέλω να σας υποβάλω σε σχέση με το μέλλον της διαχείρισης ε, αποβλήτων και φυσικά στηρίζομαι στην υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων και γι' αυτό όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει θα λάβει χώρα η πρώτη συνάντηση με τους σκιώδους σκιώδες εισηγητές για να συνεχίσουμε την πρόοδο για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και φυσικά είμαι στη διάθεση όλων των συναδέλφων εάν θέλουν να θέσουν περαιτέρω ερωτήματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φράση. για την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ιτουργκάιφ ο οποίος είναι πράγματι πολύ καλά πληροφορημένος ε, ε όπως δείχνει και το έγγραφο εργασία του. Ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για το έργο του και μας ενδιαφέρει φυσικά να υπάρχει μια προσέγγιση η οποία όπως δείχνει το έγγραφο εργασία είναι ισορροπημένη και επακριβής. Μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως τα προκατακτικά συμπεράσματα αυτής της έκθεσης, γιατί καταδεικνύουν ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη για καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας περί αποβλήτων από τα κράτη-μέλη και καλύτερη εποπτεία και αστυνόμευση της εφαρμογής των νόμων. Αυτό έχει καταδειχθεί και πρόσφατα με μια ανακοίνωση τύπου της Eurostat που κατέδειξε ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία έχει θεσπιστεί και αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάγκη της μείωσης της καταφυγής στις χωματερές και την βελτίωση σε επίπεδο ιεραρχίας αποβλήτων, δηλαδή αναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων. Συμφωνούμε επίσης ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποβλήτων και αυτή θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα για όλους μας. Κάτι ακόμα το οποίο αναγνωρίζουμε, ένα ακόμα συμπέρασμα της έκθεσης, ότι η Επιτροπή Αναφορών παίρνει ένα μεγάλο αριθμό μεμονωμένων αναφορών σε σχέση με σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Δεν είναι όλα από αυτά ε, παράνομα βέβαια η κατά της ομοθεσία, αλλά υπάρχει μια κίνηση πολιτών πολλέ φορές ότι κάπου αλλού βάλτε τα απόβλητα, δεν τα θέλω να είναι κοντά στο δικό μου σπίτι. Πιστεύουμε ότι αυτές οι αναφορές θα πρέπει με να εξεταστούν με την πρέπουσα προσοχή, αλλά θα συμφωνούσαμε περαιτέρω ότι δεν θα πρέπει να ε, παροχετεύσουν την προσοχή μας και δεν θα πρέπει να αποστρέψουν την προσοχή μας από την γενική κατεύθυνση η οποία θα πρέπει να έχει σαν στόχο μια βελτίωση γενικά της εφαρμογής και της αστυνόμευσης της νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τα συμπεράσματά σας ότι υπάρχει ανάγκη να δοθούν στην Κομισιόν οι απαραίτητοι υλικοί και ανθρώπινοι πόροι για να υπάρξει καλύτερη εποπτεία της εφαρμογής στα κράτη-μέλη και ή απαραίτητο να υπάρξει βελτίωση αυτής της εφαρμογής της νομοθεσίας περί αποβλήτων. Επομένως προσβλέπουμε στην ε, περάτωση της έκθεσής σας και την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος θέλει το λόγο? Κυρία Μέρκες. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ε, πάρα πολύ σαφή παρουσίαση των απόψεων σας σε σχέση με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι γενικά η έκθεσή σας, το έγγραφο εργασία σας περιλαμβάνει όλες τις πτυχές του θέματος. Αν θέλετε να με ρωτήσετε τι θα νόμιζα ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό το έγγραφο, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και περισσότερες αναφορές στα παραδείγματα τα οποία έχουμε δει. Έχουμε κάνει αποστολές επιτοπίως για να δούμε ορισμένες καταστάσεις. Θα ήταν χρήσιμο να περιλάβουμε και τα συμπεράσματα αυτών των αποστολών που μας δίνουν απτά παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, είχαμε την ε, αποστολή αυτή στην Καμπανία, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και αυτές οι αποστολές μας δίνουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Μήπως θα μπορούσαμε στο μέλλον, στο Pathhead ήταν αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δεύτερη που ανέφερα, μήπως θα μπορούσαμε να καταλήξουμε και σε μια σαφή διαδικασία για το πώς να αντιμετωπίζουμε αυτές τις αναφορές στο μέλλον, ώστε να ξέρουμε πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται μια αναφορά σε σχέση με την νομοθεσία φέρει αποβλήτων και πότε ξεκινάει μια τέτοια <clears throat> διαδικασία. Τι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί το έναυσμα για αυτή τη διαδικασία. Επίσης, όταν καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα, παραδείγματος χάρη, για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πάντα καλή εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος μας, με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή. Πώς θα εξασφαλίσουμε αυτό το οποίο ζητάτε εσείς στο διάλογο με τους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε λοιπόν να διαδραματίσουμε ένα ρόλο σε σχέση με το διάλογο με τους πολίτες. Μήπως θα μπορούσαμε να επιζητήσουμε με, μέσω το επιβάσει των συμπερασμάτων μας σε μια απαγόρευση για τις χωματερές ή να προτείνουμε συγκεκριμένα κίνητρα για να μειωθούν τα μη ανακυκλούμενα απόβλητα ή πώς να υποστηρίξουμε τις επαρχίες που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Πολύ καλή έκθεση. Μπορώ να υποστηρίξω όλα όσα μόλις άκουσα. Με μεγάλη χαρά άκουσα το ότι υπογραμμίζεται τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών. Οι πολίτες πρέπει να νιώθουν υπεύθυνοι αν θέλουμε να υπάρξει βελτίωση της κατάστασης και να οδηγήσουμε περισσότερους πολίτες σε περισσότερη συμμετοχή είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν παραδείγματα σαν και αυτά που αναφέρετε στην εκθεσή σας, δηλαδή ε, να δείξουμε στους πολίτες ότι όντως υπάρχει αποτέλεσμα, ότι η προσπάθειά τους ε, ε, αλλάζει κάτι, έτσι ώστε να συνεχίσουν να συμμετέχουν και να εμπλέκονται. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που είπατε. Επίσης υπάρχει και η πρόταση για μία συνάντηση με την ε, περιβαλλοντολογική υπηρεσία για τα απόβλητα. Αυτό δεν είναι απλώς ιδέα, είναι κάτι που όντως συμβαίνει. Συνεργασία με τις πόλεις οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Δηλαδή να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των ε, πόλεων, των περιοχών, που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα έτσι ώστε να υπάρξουν και λύσεις σε παρόμοια προβλήματα. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνουμε την συμμετοχή όχι μόνο πολιτών αλλά και τοπικών αρχών, περιφερειακών αρχών οι οποίες πραγματικά ενισχύονται από την γνώση και την εμπειρία άλλων. Τώρα, η ιδέα μιας νέας υπηρεσίας, δεν ξέρω αν αυτό είναι απαραίτητο. Αρκετές υπηρεσίες έχουμε. Αλλά για τα χημικά απόβλητα, παραδείγματο χάρη, μπορούμε να, απευθυνθούμε, να απευθυνθούμε στην υπηρεσία στο Ελσίνκι, όπου πραγματικά έχουν γνώση, έχουν τεχνογνωσία για χημικά ε, απόβλητα. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το όνομα αυτής της υπηρεσίας, αλλά υπάρχει και λειτουργεί στο Ελσίνκι μετά την ε, οδηγία REACH. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε τη δική τους εμπειρία για το θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντολογικά προβλήματα στην Ένωση. Ένα από τα σημαντικότερα που μας απασχολεί εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Ας δούμε λοιπόν τι άλλες προτάσεις, ιδέες μπορούμε να προτείνουμε στους πολίτες, στις αρχές σε εμά, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστούμε. Άλλοι συνάδελφοι, άλλες παρεμβάσεις. Να προσθέσω και εγώ μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την εκτιμησή μου για το έργο του συναδέλφου Τουργκάης. Βρίσκω ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική. Καλώ την ανέλαβαν οι συνάδελφοι τη Επιτροπή μα υπό το φω και του έργου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωσή της για την επικαιροποίηση της οδηγίας σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και τι παρεμβάσεις που θα χρειαστούν σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Το έργο μας στην Επιτροπή αυτή με τη στήριξη των Ευρωπαίων πολιτών μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σωστά ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πολλές αναφορές συχνά δεν έχουν ε, πραγματικές ε, βάσεις και αιτιολογίες. Ε, πιθανό αυτό. Γι' αυτό εξαντλούμε όμως κάποιες περιπτώσεις και στεκόμαστε σε αναφορές όπου μέσω των καταγγελιών που φτάνουν στην Επιτροπή μας βλέπουν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, κρίσιμα προβλήματα. Έτσι λοιπόν έργο των πολιτών μπορεί να θεωρηθεί και αυτό και αυτό το έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συνεχή έλεγχο και την παρακολούθηση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας των συνθηκών θα πρέπει να ενεργεί καθημερινά. Οι αναφορές είναι μικρά, μικρές ευκαιρίες να επικεντρωθούμε σε λεπτομέρειες της υλοποίησης των κοινοτικών οδηγιών. Η ενίσχυση λοιπόν της συνεργασίας είναι σημαντική τα συμπεράσματα που αναφέρονται σε διάλογο με τους Ευρωπαίους πολίτες, με τους πληθυσμούς, είναι πολύ εύστοχα. Ο διάλογος με τους πολίτες, μέσω της δικής μας της Επιτροπής, μπορεί πράγματι να αξιοποιηθεί ώστε και η Εκτελεστική Επιτροπή ε, να φέρει πέρα στην αρμοδιότητα αυτή που της αναλογεί. Και έναν αντιασμό έχω στο σημείο 36 σε σχέση με την επαναθεώρηση της ε, διανομής των κονδυλίων, της κατανομής μάλλον των κονδυλίων και το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ε, κονδύλια του Ταμείου Συνεχής για θέματα περιβάλλοντος και για διαφορετικά ζητήματα. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και σε σχέση με όσα συζητάει η Επιτροπή Περιφερικής Ανάπτυξης για τη χρησιμότητα και το εύστοχο μιας τέτοιας ε, αλλαγής όπως αντιτυπώνεται στα συμπεράσματά μας. Θεωρώ ότι το έργο είναι αυτό για το χρονοδιάγραμμα. Έχω δώσει ήδη τα σημαντικότερα χρονικά σημεία. Τα έχει πει και ο συνάδελφος Ιτρουγκάης. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για τα συμπεράσματά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από το τέλος αυτά που είπε η Πρόεδρος ότι είναι σημαντικό το έργο. Όχι μόνο σημαντικό αλλά είναι ένα απαραίτητο έργο γιατί είναι γεγονός ότι υπήρξαν πάρα πολλέ αναφορέ οι οποίες φτάνανε στην Επιτροπή μας σε σχέση με τα θέματα περιβάλλοντος και εμεί θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε συνέχεια. Υπήρξε, υπήρχε ένα είδος νησίδος ακινησίας στην Επιτροπή μας στο παρελθόν έναντι όλων αυτών των αναφορών που ερχόντουσαν σε σχέση με τα απόβλητα. Γι' αυτό θα ευχαριστήσω και την εκπρόσωπο τη Κομισιόν που υποστηρίζει τα προσωρινά αυτά συμπεράσματα, γιατί αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας να υπάρξει και μια συμπληρωματικότητα εργασία μεταξύ της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τόσες ε, αναφορές οι οποίες έχουν φτάσει για τα θέματα των αποβλήτων και όπως τόνισε και η Πρόεδρός μας νομίζω ότι εδώ γίνεται με τρόπο ακριβή και εμπεριστατωμένο μια εργασία για να αντιμετωπίσουμε τις τεκμηριωμένες αναφορές οι οποίες έρχονται στην Επιτροπή μας. Βέβαια μπορεί και η Γραμματεία να σας πει ότι έρχονται πάρα πολλές αναφορές, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε να προωθήσουμε τις αναφορές οι οποίες έχουν τεκμηριωμένο χαρακτήρα, ώστε να αντιμετωπιστούν με τον απαραίτητο εμπεριστατωμένο τρόπο. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να πω είναι καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μέρκης και την κυρία Άουκεν για τα καλά τους λόγια. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα αυτό το οποίο είπε η κυρία Μέρκης, στην οποία την πέρα. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσατε να κάνετε πολύ καλό έργο σας και όδηση συγγήτρια όπως και η κυρία Άουκεν για μια διαδικασία η οποία θα εξασφαλίσει ότι όταν φτάνουν οι αναφορές να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης. Όπως είπα και προηγουμένως, νομίζω ότι όπως έκανε και με την έκθεση της κυρίας Άουκεν για την ε, τα οικιστικά θέματα, όπου και εκεί θα έρθουν και άλλες ε, αναφορές, θα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να κατανέμουμε τις εκθέσεις μεταξύ των διαφόρων εκθέσεων. Μπορούμε να κρατήσουμε πάντα αποφάσεις οι οποίες είναι σαφείς. Αποφάσεις οι οποίες έχουν και κάποια εχμηρότητα. Να ξέρουν οι πολίτες ότι μπορούν δηλαδή να απευθυνθούν στην δική μας Επιτροπή και ο οποιοδήποτε ο οποίος κάνει μια αναφορά να ξέρει ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων πολίτων σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Τώρα η κυρία Μέρκης και η κυρία Άουκεν συμφωνήσαμε στο ότι θα μπορούσαμε να θέτουμε στο έγγραφο αυτό, στην έκθεση αυτή, παραδείγματα Ελπίζω να μην καταλήξουμε όμως σε τοπικιστικές αντιμετωπίσεις, γιατί αυτή είναι μια έκθεση η οποία πρέπει να καλύψει όλη την Ευρώπη. Όλους τους Ευρωπαίους πολίτες πρέπει να είναι μια έκθεση η οποία θα έχει εγκυρότητα και για ένα Δανό, για ένα Εστονό, για ένα Ιταλό, για ένα Βρετανό και όχι να λέμε ότι εδώ είναι αυτό ή εδώ δεν έγινε εκείνο να έχουμε μια ευρύτερη λοιπόν αντιμετώπιση για το παρόν και για το μέλλον, για το πώς θα πρέπει να επιληθούν προβλήματα αυτά και τώρα φυσικά αν υπάρχουν καταφανή παραδείγματα, χτυπητά παραδείγματα, μπορούμε σίγουρα να τα συμπεριλάβουμε στην έκθεση αυτού του είδους. Η κυρία Άουκεν αναφέρθηκε και στο θέμα της επαφής με τους πολίτες. Σύμφωνο και το έχω τονίσει αυτό στο έγγραφο εργασίας, και σίγουρα μπορούμε να δώσουμε μια πιο στεναρή διατύπωση σε σχέση με την <clears throat> επαφή με τους πολίτες. Μια ακόμα ιδέα που νομίζω ότι προέκυψε με αυτά που συζητήσαμε την κυρία Άουκεν, να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία των πολιτών μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, γιατί θα μπορούσε να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα η παρέμβαση πολιτών από διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα αλλά ελπίζω ότι εσείς θα την επεξεργαστείτε λίγο περισσότερο για να μπορέσετε να μας δώσετε μια σαφέστερη διατύπωση ώστε να τη συμπεριλάβουμε στο, έκθεση, στο έγγραφο αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα, αν μπορείτε εσείς να μας παρουσιάσετε μια πιο συγκεκριμένη, μια πιο εκτενή ε, διατύπωση για τα θέματα αυτά. Δεν σας το ζητάω τώρα να το κάνετε, αλλά νομίζω ότι στη συνέχεια της συζήτησης θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο και θα μπορέσετε να μας δώσετε και μερικές σκέψεις δικές σας σε σχέση με το θέμα αυτό. Και για να κλείσω, είπε η κυρία Άουκεν ότι έχει αμφιβολίες για τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας, ενός νέου αποκεντρωμένου φορέως. Γιατί αναφέρθηκε αυτό από ό,τι γνωρίζω για εσάς κύριε Άουκεν, συμφωνείτε στο ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται να έχουμε περαιτέρω αποκεντρωμένους φορείς, αλλά να εργάζονται οι φορείς οι οποίοι υπάρχουν σε πιο αποτελεσματικό, με πιο αποτελεσματικό τρόπο και να δίνουν λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, δηλαδή να δίνουν απαντήσεις στους πολίτες. Πολλές φορές ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε είναι ότι δημιουργούμε πάρα πολλά εισιτούτα, πάρα πολλούς αποκεντρωμένους φορείς και όλα αυτά. Στη συνέχεια όμως είναι απογυμνωμένοι αυτή η φορείς από περιεχόμενο και από απαντήσεις στις πραγματικές ερωτήσεις και τα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν ξέρω λοιπόν αν το θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερους ή λιγότερους αποκεντρωμένους φορείς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι φορείς οι οποίοι είναι εν υπάρξει που υπάρχουν να μπουν στο παιχνίδι της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίσουμε ως Επιτροπή Αναφορών και που επανέρχονται συνέχεια στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Άουκε νομίζω θέλει να πει κάτι. Ναι, για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Δεν έλεγα απλώ συνεργασία μεταξύ πολιτών ότι πρέπει να προωθήσουμε, αλλά και μεταξύ των αρχών. Αυτό δεν είναι απλώς ε, ιδέα που υποβάλλω, αλλά κάτι που πραγματικά στηρίζεται στην εμπειρία μας στην Κοπενχάγη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εμπνευστούμε από αυτό που έγινε, να μας δώσουν μάλιστα και τη διατύπωση. Δεν είναι απλώς συμμετοχή πολιτών, δεν προσπαθώ να δημιουργήσω ένα μη κυβερνητικό οργανισμό, αλλά συνεργασία αρχών. Και αυτό πρέπει να υποβάλουμε εδώ σαν ιδέα. Αλλά και η Eurostat, η οποία με θεαματικό τρόπο έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τομέα της στατιστικής. Όντως, τα πράγματα σήμερα είναι διαφορετικά και εάν δεν αναφέρουμε αυτά τα παραδείγματα, όλη αυτή η καταπληκτική δουλειά που έχει γίνει, η οποία πολλές φορές δεν βγαίνει προς τα έξω, θα χαθεί. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όλα αυτά είναι χρήσιμα, ότι η δουλειά που κάνουμε εδώ είναι χρήσιμη και να δώσουμε, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία αποδεικνύουν στον κόσμο ότι γίνεται καλή δουλειά και ότι και εμείς κάτι κάνουμε. Γι' αυτό και στήριξα την πρόταση της Τζούδιθ όσον αφορά αυτό που και εσείς εξάλλου αναφέρατε. Στο τέλος του μήνα πάμε στη Βουλγαρία να δούμε ότι υπάρχει περιπτώση υπάρχει αποτέλεσμα στη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες και οι φορείς που υπάρχουν δεν έχουν περιεχόμενο δεν έχω στοιχεία για να το πω αυτό έτσι. Είναι ίσως λίγο γενικευμένο αυτό σαν ιδέα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αντίθετα να επιμείνουμε λίγο παραπάνω στα παραδείγματα και στα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ζητά κανεί το λόγο. Να κλείσουμε λοιπόν τη συζήτηση για το θέμα αυτό και να περάσουμε στο επόμενο σημείο 8 αναφορά αριθμός 16-17 το 2009 για το πρόβλημα του λατομείου ασβεστόλιθου Σόμντε Λαμπριζερή στην Λακουρών τη Σαρόντ από δύο κοιτάσματα υπογείων υδάτων. Το λόγο έχει ο κύριος Μάρτιν λοιπόν, στον οποίο δίνω το λόγο για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές. Εκπροσωπώ εδώ τους πολίτες που ζουν γύρω από αυτό το λατομείο. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν την αναφορά 16-17 του 2009 και θα καταγγείλω την άδεια για την εμβάθυνση αυτού του λατομείου που βρίσκεται στην Γαλλία. Η παρουσίασή μου έχει δύο τμήματα. Καταρχήν θα ήθελα να σας πενθυμίσω την άδεια αυτή που εδόθη για την εκμετάλλευση αυτού του λατομείου και δεύτερον ποια είναι τα σημεία τα οποία καταγγέλουμε γιατί θεωρούμε ότι παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο και την οδηγία. Πρόκειται για ένα λατομείο που βρίσκεται στη Γαλλία, στο διαμέρισμα της Σαρόντ. Πρόκειται για την εταιρεία Lafarge Cimento που εκμεταλλεύεται αυτό το λατομείο εδώ και πολλά χρόνια και έχει γίνει αποδεκτό από τους πολίτες. Σήμερα όμως δεν μπορεί πλέον να επεκταθεί σε επιφάνεια αυτό το λατομείο. Ζήτησαν λοιπόν έκαναν μια πρώτη αίτηση για το διαμέρισμα να υπάρξει επέκταση εις βάθος αυτού του λατομείου. Δηλαδή θα πρέπει να διαπεραστούν δύο κοιτάσματα υπόγειων υδάτων, κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκχυθούν τα ύδατα αυτά από τα κοιτάσματα τα οποία θα αποξηρανθούν. Εμείς ε, αμφισβητούμε μια σειρά σημείων τα οποία θα σας παρουσιάσω. Εδώ βλέπετε το λατομείο με τις επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος. Βλέπετε τα δύο ποτάμια, ένα στο βορρά και ένα στο νότο, που θα χρησιμοποιηθούν για να εκχυθούν τα ύδατα όταν υπάρξει αυτή η επέκταση εις βάθος του λατομείου. Υπάρχει και η περιοχή η οποία έχει ταξινομηθεί στο Natura 2000 καθώς και οι πηγές οι οποίες και αυτές θα αποξηρανθούν. Πρόκειται λοιπόν για μια επέκταση της τάξης των 35 μέτρων. Θα φτάσουμε δηλαδή στα 25 μέτρα και θα διαπεραστούν δύο κοιτάσματα υπόγειων υδάτων την ίδια ώρα. Τα κοιτάσματα αυτά θα ρηπανθούν και τα ύδατά τους τα οποία θα ξεπεράσουν τα 2,6 εκατομμύρια κυβικά νερού, κάτι το οποίο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μια πόλη 50.000 κατοίκων. Εδώ βλέπετε και την τομή του λατομείου με το σημερινό επίπεδο. Βλέπετε στην πράσινη γραμμή το σημερινό επίπεδο και την πρόταση για επέκταση του λατομείου εις βάθος. Βλέπετε επίσης τα ύδατα τα οποία θα εκχυθούν στην λεκάνη του λατομείου με τη δημιουργία ενός μικρού ποταμού. Βλέπετε επίσης τα χαρακτηριστικά, τα φυσικά χαρακτηριστικά των υδάτων αυτών. Θεωρούμε ότι η άδεια αυτή δεν είναι συμβατή συγκεκριμένα με την ε, Οδηγία Πλαίσιο 2060, παράγραφος 4, άρθρο 4, παράγραφος 1, συγγνώμη, που αναφέρεται στην ε, επιδίνωση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων και βεβαίως τις επιπτώσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος. Σήμερα ξέρουμε ότι η περιοχή αυτή ήδη γνωρίζει ξηρασία. Την προηγούμενη εβδομάδα ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφτηκε την περιοχή μας και δήλωσε συγκεκριμένα μέτρα κατά της ξηρασίας. Επίσης, άρθρο 4, σημείο Β καθώς και το παράρτημα 5 που αναφέρεται στην καλή κατάσταση όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα των υδάτων αυτών. Σήμερα τα κριτήρια αυτά δεν εκπληρούνται ούτε όσον αφορά την ποσότητα, ούτε όσον αφορά τη μείωση του επίπεδου και της ε, ποιότητας των υδάτων αυτών στα κοιτάσματα υπογείων υδάτων. Αυτό θα έχει επιπτώσεις σε μία περιοχή που ξεπερνάει τα 2 χιλιόμετρα γύρω από το λατομείο. Επίσης, στο παράρτημα 5 βλέπουμε ότι υπάρχουν οι αξίες που έχουν καθοριστεί από τις γαλλικές αρχές και οι οποίες δεν τηρούνται όσον αφορά τουλάχιστον τη χημική ποιότητα των υδάτων αυτών, όσον αφορά το pH, εδώ υπάρχει μία ψαλίδα 5 6,5 έως 8,5. Σήμερα βλέπουμε ότι το pH των υδάτων αυτών έχει ξεπεράσει το 7,3. Η ύψιστη επίσης θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμοί. Σήμερα βλέπουμε ότι το φυσικό περιβάλλον δεν ξεπερνά τους 15 βαθμούς. Επίσης υπάρχουν και διάφορες άλλες ουσίες που ξεπερνούν τις προβλεπόμενες ανώτατες αξίες, όπως παραδείγματο χάρη τα έλαια εδώ προβλέπεται να ηχηθούν πάνω από 100 λίτρα έλαιο ανά 24 ώρο, κάτι που ξεπερνάει κατά πολύ την ποιότητα των υδάτων αυτών. Αναφέρομαι επίσης και στην οδηγία του 2060, οδηγία πλαίσιο, και θεωρούμε ότι η συχνότητα δεν ε, τηρείται. Εδώ βλέπουμε ότι η οδηγία πλαίσιο προβλέπει πολύ χαμηλότερες ανώτατες αξίες. Η ποιότητα των υπόγειων υδάτων επίσης, τα υπόγεια οικοσυστήματα. Βλέπουμε ότι η εμβάθυνση αυτού του λατομείου θα έχει επιπτώσεις σε όλες τις ε, γύρω περιοχές, της στα υπόγεια ύδατα που περιβάλλουν αυτό το λατομείο. Θα υπάρξει λοιπόν σύρανση, εξαφάνιση των χερσαίων οικοσυστημάτων και προστατευμένων ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα 2 και στο παράρτημα 4 της οδηγίας για την χλωρίδα και την πανίδα, χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία άδεια για την καταστροφή αυτών των ειδών. Τέλος, όσον αφορά την οδηγία 2006-118 κατά της ρήπανσης των υπόγειων υδάτων, υπάρχουν εδώ διαφορετικές μετρήσεις όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτών των υδάτων, αλλά και μία υποβάθμιση της ποιότητας των ε, υδάτων αυτών. Το 2007 διαβάσαμε στον ε, τύπο ότι μία έκχυση διαφόρων ουσιών ήδη μόλυναν τα γύρω ποτάμια και προκάλεσαν θνησιμότητα των ψαριών. Επίσης, οδηγία του 2001-42 χωρίς να υπάρξει απολύτως καμία συγκεκριμένη παρουσίαση στοιχείων για την υποκατάσταση αυτών των ειδών και καμία μελέτη αντικτύπου όσον αφορά το περιβάλλον. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία είναι πλούσια σε άργυλο, δεν υπάρχει εδώ καμία μελέτη για την αντίσταση και την ανθεκτικότητα του εδάφους. Καμία μελέτη δεν έχει γίνει και καμία απάντηση δεν έχει δοθεί από τις γαλλικές αρχές. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ σημαντικές επί του περιβάλλοντος, εξαφάνιση πόρων, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές κατοίκων. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη σε όλα αυτά τα στοιχεία και ζητούμε από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρέμβει προς τις γαλλικές αρχές έτσι ώστε να αναθεωρηθεί όλο αυτό το έργο και να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις και να μην υπάρξει αυτή η επέκταση εις βάθος του λατομείου με συγκεκριμένες ε, επιπτώσεις όπως σας παρουσίασα και για τα υπόγεια ύδατα αλλά και για τους μέλλοντες κατοίκους της περιοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ με εξαιρετική παρουσίασή σας από την Επιτροπή κυρία Μπράντμαρκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον αναφερόμενο για όλες τις πολύ συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά αυτή την αναφορά που μας παρουσιάζει σήμερα Όντως πρόκειται για θέματα που αφορούν την οδηγία πλαίσιο και τα υπόγεια ύδατα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποσότητα, την ρήπανση των υπόγειων υδάτων, αλλά και τις επιπτώσεις επί των οικοσυστημάτων και των υδάτων επιφανείας. Η Επιτροπή σήμερα μπορεί να λάβει υπόψη της όλα αυτά τα επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία πολύ συγκεκριμένα μας ενημερώνουν για το ποιες διατάξεις της οδηγίας ενδεχομένως παραβιάζονται. Μπορούμε λοιπόν να αξιολογήσουμε καλύτερα εάν και εφόσον αυτή η άδεια έχει λάβει υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο αλλά και της αντίστοιχης οδηγίας 2006-118. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπελάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τη στιγμή που είδα ότι πρόκειται εδώ για το θέμα Λαφάρτζ, εγώ προτιμήσα να ολοκληρωθεί το θέμα, η αναφορά αυτή, διότι από τη στιγμή που έγινε η προσφυγή, πριν μάλλον γίνει η προσφυγή, είδαμε ότι οι δημοτικές αρχές είχαν ταχθεί υπέρ του προγράμματος Λαφάζ. Από τον αναφερόμενο όμως ακούμε ότι η προσφυγή φαίνεται να είναι σωστά αιτιολογημένη και θεμελιωμένη. Οπότε, αν δεν θέλουμε να παρεμβληθούμε σε μια διαδικασία που νομίζω ότι εκδικάζεται σε εθνικό επίπεδο, καλό θα ήταν να αφήσουμε ανοιχτό το ζήτημα της αναφοράς αυτής. Ώστε προηγουμένως η Δημοτική Αρχή να τοποθετηθεί το ίδιο και σε εθνικό επίπεδο και να δούμε κατά πόσο υπάρχει σεβασμός ή όχι της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Υπήρξε μια μελέτη η οποία είχε επίσης δώσει θετική αποτίμηση και στον όλο, στο όλο ντοσιέ και το δίκτυο Transnatura για το περιβάλλον ήταν υπέρ του όλου προγράμματος, όπως και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι στην αρχή δεν υπήρχε πρόβλημα παραβίασης των ευρωπαϊκών οδηγιών. Τέλος, θυμίζω απλώς ότι η προσφυγή που πρόσφατα υποβλήθηκε δεν είναι ανασταλτικού χαρακτήρα. Ας αφήσουμε λοιπόν σε κρεμότητα αυτήν την αναφορά, ώστε να ολοκληρωθεί το ντοσιέ ανάλογα με την εκδίκαση της προσφυγής. Και έπειτα και εμείς στην Επιτροπή Αναφορών θα μπορούμε να τηρήσουμε μια συγκεκριμένη στάση. Άλλες παρεμβάσεις. Όχι. Ο αναφερόμενος θέλει να προσθέσει κάτι βάσει των όσων άκουσε. Μια κλασική διαδικασία έγκριση στην ε, Γαλλία. Τώρα μπορεί μέσα στα πλαίσια αυτά να υπάρχουν στοιχεία τα οποία αφορούν ελλείψεις και λαθασμένες ενέργειες. Έχει φτάσει όμως τώρα η διαδικασία αυτή ενώπιον των αρχών. Η μόνη προσφυγή η οποία εκκρεμεί είναι μια καθαρά διοικητικού χαρακτήρα ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα πρέπει να γίνει γνωστό πολύ σύντομα. Η προσφυγή λοιπόν η οποία αφορά εδώ την ε, συνάφεια με τις ευρωπαϊκές οδηγίες μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και εμείς από την πλευρά της δικής μας ε, ε Ένωσης και μέσα από την ε, τεκμηρίωση που έχουμε δώσει έχουμε ζητήσει να υπάρξει μια σε εξέταση των πραγματικών γεγονότων που συνάπτονται με αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Άρα ε, υπάρχει εδώ ένα αίτημα να παραμείνει ανοιχτό το ζήτημα της εν λόγω αναφοράς. Σκόπιμο θα ήταν, όχι μόνο για να αναμένουμε και την εκδίκαση της ε, υπόθεσης από τις διοικητικές αρχές της Γαλλίας, αλλά για να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια επιπλέον αποτίμηση του θέματος βάσει των στοιχείων που σήμερα μας προσκόμισε ο αναφερόμενος. Ήταν η παρουσίασή του ιδιαίτερα περιστατωμένη, πολύ λεπτομερής και δεδομένης και της τελευταίας ε, Ε, τοποθέτησης της Επιτροπής που έλεγε ότι θα αποφανθεί επί των προσκομιστέντων στοιχείων. Σήμερα έχουμε και άλλα που προσκομίστηκαν, οπότε καλό θα ήταν να τα λάβετε και αυτά υπόψη σας. Ζητώ λοιπόν και από τον συνάδελφο Μπουλάν και από τον αναφερόμενο να παρακολουθήσουν την τοπική εκδίκαση του όλου θέματος ώστε να λάβουμε κι εμείς γνώση για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας. Παραμένει λοιπόν ανοιχτό το θέμα της αναφοράς. Ευχαριστώ τον κύριο Μάρτιν για την παρουσία του εδώ και περνούμε στις αναφορές που περιλαμβάνονται από το σημείο 9.331 του 2010 από τον κύριο Ιγνάσιο Ρου Υπέρες Αρέγκουι για την κατάσταση των ελεγκτών αναέρειας κυκλοφορία στην Ισπανία και το ίδιο και την αναφορά 651 του 2010 που υπέβαλε ο Χουάν Μαρία Γκαρθία Ζιλ. Η δεύτερη αναφορά συγκεκριμένα αναφέρεται στις συνδικαλιστικές ενώσεις των ελεγκτών. Είναι παρόντες και οι δύο αναφερόμενοι, οπότε να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Γνάσιο Ριπέρες Αρέγκουι. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, μέλη του Προεδρείου, μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσω την άποψή μου ενώπιόν σας. Στις 5 Φεβρουαρίου του 2010 η Ισπανική κυβέρνηση άλλαξε δραστικά την ε, νομοθεσία σε σχέση με τον εναέριο έλεγχο. Αυτή η αλλαγή σημαίνει μια πραγματικά επιταγή εν λευκό για να αλλάξει και η εφαρμογή της νομοθεσίας για τους εναέριους ελεγκτές. Μία αύξηση επομένως 60% του φόρτου εργασίας μας τα επόμενα χρόνια. Αυτή η αύξηση γίνεται χωρίς να υπάρξει κάποιος έλεγχος της ικανότητάς μας να φέρουμε σε πέρα στο έργο του ενάριου ελεγκτή κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία μελέτη ασφάλειας σε σχέση με την δυνατότητα να συνεχίσει το έργο των ενάριων ελεγκτών κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αυτή η αλλαγή ακυρώνει όλα αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής από το 1992 μετά από συλλογικές διαπραγματεύσεις πριν από 20 χρόνια περίπου. Ο στόχος από την πλευρά των αρχών είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αρχών εναερίου ελέγχου στην Ισπανία. Παρ' όλα αυτά, μετά από 16 μήνες, κατά τους οποίους λειτουργεί αυτό το νέο εργασιακό και ε, ρυθμιστικό πλαίσιο, δεν υπήρξε καμία αλλαγή της ε, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της εργασίας. Υπήρξε μια αξιοσημείωτη αύξηση των εργασιακών συγκρούσεων Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα των ε, εναρίων ελαγκτών που έχουν ιατρικά και ιδίως ψυχιατρικά προβλήματα. Υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στους ε, ισπανικούς εθέρες οι οποίες έχουν ε, αναφέρει προβλήματα. Παραδείγματος χάρη το έτος 2009 η καθυστέρηση η συνολική καθυστέρηση έφτασε τις 900.000 ε, λεπτά καθυστέρησης. Μέσα στο νέο πλαίσιο του 2010 έφτασε στα 5 εκατομμύρια λεπτά ε, καθυστέρησης. Τι έγινε λοιπόν για να υπάρξει μια τόσο μεγάλη, πέντε φορές μεγαλύτερη συνολική καθυστέρηση. Και επίσης υπήρξε και ένας πάρα πολύ ανησυχητικός αριθμός επεισοδίων σε ε, επίπεδο ενέργειας κυκλοφορίας βάσει και των στοιχείων της Eurocontrol. Βάσει των στοιχείων αυτό το 2010 στην Ισπανία υπήρξε αύξηση 96% των συνολικών εναέριων επεισοδίων πάνω από τους εθέρες της Ισπανίας. Με μια απλή σύγκριση ο... οι εθέρες του Ηνωμένου Βασιλείου όταν λέμε, όταν λέμε για επεισόδια, υπάρχουν επεισόδια κατηγορίας α, β, γ, δ κτλ. Α σημαίνει σχεδόν σύγκρουση εν πτήση δύο αεροσκαφών. Στους ε, Βρετανικούς εθέρες το 2010 είχαμε 2.100 2.100.000 κινήσεις αεροσκαφών και δεν υπήρξαν καθόλου επεισόδια τύπου α, τύπου β. Βλέπετε λοιπόν ότι στην, ε, επίσης στη Γερμανία με 2.700.000 κινήσεις, 4 επεισόδια τύπου Α και 3 επεισόδια τύπου Β. Και τώρα για την Ισπανία. Στην Ισπανία το 2007-2010 είχαμε με 1.700.000 κινήσεις αεροσκαφών είχαμε επεισόδια τύπου Α σχεδόν συγκρούσεις όπου οι πιλότοι αναγκάστηκαν να κάνουν χειρισμούς τελευταία στιγμή για να αποφύγουν τις συγκρούσεις 47 επεισόδια τύπου Α και 92 τύπου Β. 47 επεισόδια στο, σε ένα χρόνο, δηλαδή τέσσερις φορές το μήνα υπήρχε ένα τέτοιο επεισόδιο, σχεδόν κάθε εβδομάδα υπήρχε ένα τέτοιο επεισόδιο. Μια φορά λοιπόν κάθε εβδομάδα δύο αεροπλάνα θα μπορούσαν να είχαν συγκρουστεί στον Ισπανικό εναέριο χώρο. 47 Ιωνί συγκρούσεις λοιπόν. Αν σκεφτείτε ότι κάθε αεροπλάνο έχει περίπου 200 επιβάτες, περίπου 20.000 Ευρωπαίοι και μη Ευρωπαίοι χρήστες του Ισπανικού ενάριου χώρου πέρασαν παρατρίχα από μια ενάρια καταστροφή. Αν το δούμε λοιπόν συνολικά το θέμα αυτό, τα αποτελέσματα αυτών των δραστικών αλλαγών που επιφέρθησαν στον ενάριο έλεγχο ήταν πραγματικά δραματικά. Δεν υπάρχει σεβασμός στην Ισπανία της οδηγίας για, τον, για την εναέρια ασφάλεια, ούτε καν και η οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Και τώρα, ζητώ συγγνώμη και από τους μεταφραστές, θα σας κάνω μία απαρίθμηση όλων των συνθηκών που δεν τηρούνται. Ξεκινώ με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Λισαβόνης. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα. Κανονισμός 2096 κάθετος 2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να τονίσω ότι στον κανονισμό αυτό υπάρχει μια δεσμευτικότητα για όλους αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας για να εξασφαλιστεί η ύπαρξη ενός συστήματος ασφαλείας που μπορεί να διαπιστώσει όλους τους λειτουργικούς κινδύνους και που θα πρέπει να έχει ένα υποχρεωτικό χαρακτήρα και να υπάρξει υποχρεωτικό έλεγχο πριν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στον ενέργειο έλεγχο. Θα πρέπει λοιπόν να ερευνηθεί και να προσωμιωθεί όποια, το αποτέλεσμα οποιασδήποτε διαδικασία. Στην Ισπανία αυτό δεν γίνεται. Κανονισμός 1989-31, ε, η οδηγία 1989 κάτω 791 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Οδηγία 98 κάτω 59, η Οδηγία 2003 κάτω 88 Ευρωπαϊκή Ένωση, η Οδηγία 2002 κάτω 14 Ευρωπαϊκή Ένωση, η 2000 κάτω 78 Ευρωπαϊκή Ένωση, 1999 κάθετο 70 του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να τονίσω και πάλι σε αυτή την οδηγία γιατί έχει να κάνει με το σχέδιο, με την συμφωνία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων και Εργοδοτών και πάλι μιλάω για τους συλλογικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τα συνδικάτα στις δημόσιες ε, επιχειρήσεις δεν είναι συμβατά όλα αυτά με τις ε, ε, αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού ε, πολιτικής αεροπορίας ούτε και με τις ε, ρήτρε του Eurocontrol για την εναλλαγή των ε, βαρδιών στους εναέριους ελεγκτές. Παραβιάζεται επίσης μία σειρά από ρυθμίσεις των, των εργαζομένων για τους το, εργαζόμενους στον τομέα μεταφορών, για τους πιλότους οι οποίοι εργάζονται στις εναέριες μεταφορές Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν συμμετάσχει στην έρευνα που ζητήσατε ως Επιτροπή Αναφορών να κάνουμε. Το νέο αυτό πλαίσιο, χωρίς διάλογο, επιβάλλει στους ε, ενάριους ελεγκτές να δεχτούν το νέο πλαίσιο. Υπήρξαν πάνω από 1.300 αναφορές και πάνω από 10.000 υπογραφές συλλέχθησαν από Ευρωπαίους πολίτες που ζητάμε τα εξής. Πρώτον, να επαναφερθεί η νομιμότητα σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους Ισπανούς ενάριους ελεγκτές. Να επαναφερθεί η ευρωπαϊκή νομιμότητα. Να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τον ε, χώρο αυτοεργασίας μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ενέου χώρου. Να υπάρξουν οι απαραίτητε μελέτες για θέματα ασφάλειας και διαπίστωση λειτουργικών κινδύνων προτού, προτού εφαρμοστεί οποιαδήποτε μεταρρύθμιση η οποία μπορεί να επηρεάσει το σύστημα του εναέριου ελέγχου. Τέλος, ζητούμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει πέρας στο καθεστώς το οποίο υφίστανται οι Ισπανοί εναέριοι ελεγκτές οι οποίοι εργάζονται μέσα σε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο δεν μπορεί να υπάρξει εξασφάλιση της εναέριας ασφάλειας. Πάνω από τέσσερις από 400 ε, ελεγκτές έχουν, έχουν απολυθεί και έχουν αντιμετωπίσει διοικητικά, πειθαρχικά και ποινικά μέτρα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν παρενόχλησης και καταστροφής της ασφάλειας έχει διαπιστωθεί και από την Διεθνή ε, ε, Ένωση ΦΑΤΚΑ η οποία έχει ζητήσει να αποβληθεί η Ισπανία από τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες. 4 Δεκεμβρίου του 2010 έλαβε χώρα ένα γεγονός χωρίς προηγούμενο. Οι, Οι εθνικές αρχές με ένοπλες συνοδείες υποχρέωσαν τους ε, ενέργειους ελεγκτές να φέρουν σε πέρα στο καθήκον τους υπό καθεστώς ε, εξαναγκασμού. Αυτό είναι κατά όλων των ε, των κανόνων της Eurocontrol και των ενιαίων εθέρων. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τις ευρωπαϊκές αρχές και χαίρομαι γιατί οι, τα, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται κοντά στους πολίτες και μας δίνουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την ε, ε, αναφορά μας σε εσάς. Ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει ο κυρίος Αντάρτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Εξ ονόματος του, της Ένωσης των ε, Ισπανών Ενέαριων Ελεκτών που εκπροσωπεί το συνδικάτο μας το ΟΥΣΚΑ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω την άποψή μας. Όπως έλεγε και ο συνάδελφός μου θα μπω κατευθείαν στην ουσία του θέματος. Η κατάσταση αυτή ε, είναι πάρα πολύ σοβαρή, αλλά δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Στις 5 Φεβρουαρίου 2010, μετά από την ε, δράση της ΑΕΝΑ, που είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι εργοδότες μας, ε, ανέφεραν ότι μονομερώς καταγγέλνουν τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας νέας συλλογικής συμφωνίας, η Ισπανική κυβέρνηση, προτάσει του Υπουργείου Ανάπτυξης, ε, διετύπωσε ένα βασιλικό διάταγμα για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο εναέριου ελέγχου και τελικά αντικαταστάθηκε από τον νόμο 2009-2010 του 14 Απριλίου. Όλες αυτές οι νομικές Διατυπώσει βασίζονται σε ορισμένα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία κατέδειξαν ενώπιον τη κοινή γνώμη και ενώπιον του Ισπανικού Κοινοβουλίου ότι πράγματι ήταν αυτά τα οποία υποστήριζαμε εμεί ω εναέρια διαλεκτές και όχι αυτά που υποστήριξε η Ισπανική κυβέρνηση. Η περιορισμένη ε, παραγωγικότητα η οποία μας καταγγέλλεται βασίζεται στα λαθασμένα, στα στρεβλά στοιχεία τα οποία έχει δώσει η ΑΕΝΑ τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τον αριθμό των ελεκτών που είναι εν υπηρεσία. Όταν περιλαμβάνει όλους τους ελεκτές, ακόμα και αυτούς οι οποίοι είναι στον τομέα του σχεδιασμού και της, διοικη... και του... και της διοίκησης, δεν οδηγεί αυτό σε σαφή στοιχεία σε σχέση με την παραγωγικότητα των εναερίων ελεκτών, που είναι πολύ έτσι μικρότερα της πραγματικότητας. Αν χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα της Eurocontrol, θα αυξηθεί αυτή η παραγωγικότητα σε κατά 30% και θα φτάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τονίστηκε και από τους βουλευτές του, των Κόρτες στην, ε, στην Ισπανική Βουλή και η ΑΕΝΑ παρεδέχθη ότι ήταν λαθασμένες οι πληροφορίες που είχαν αποστείλει. Κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό είναι το γεγονό ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εκστρατεία στον τύπο για να τονίσει ότι, ότι εργαζόμαστε λιγότερο από οποιονδήποτε στην Ευρώπη. Από όλου του ενέργειου ελεκτέ. Το Eurocontrol όμω έχει σαφεί πληροφορίε για τα θέματα αυτά. Το προήμιο του της ε, συμφωνίας της, ε, του κανονισμού που έχει γίνει σε σχέση με τα θέματα αυτά αναφέρεται και αναφέρει και το εργαζόμαστε εμείς περισσότερο από οποιοδήποτε άλλου ενεργούς ελεκτές στην Ευρώπη. Και αυτό έχει δημοσιευτεί και έχω εδώ τις ε, ε, μαρτυρίες που έχουν καταθέσει σε σχέση με το θέμα αυτό. Παρά αυτές λοιπόν τις αλλαγές που ήταν σημαντικές, και βασιζόμενοι στα προηγούμενα δύο στιμία που ανέφερα, τους τελευταίους μήνες η Ισπανική κυβέρνηση έχει εκδώσει 27 διατάγματα, νόμους ή εγκύκλειους υπουργικές, βάσει των οποίων συνεχίζει την προσπάθειά του να τροποποιήσει άρδιν το πλαίσιο το εργασιακού μας όλα αυτά συγχρόνως με μια εκστατεία στα μέσα ενημέρωσης, στην οποία μας κατηγόρησαν ότι είμαστε εκβιαστές, ότι είμαστε απαγωγείς, ότι είμαστε κλέφτες κτλ. Η πρόσφατη έγκριση στις 9 Μαρτίου του νέου πλαισίου αυτού που αναφέρθηκαν σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες των εναρίων ελεγκτών δεν έχει επιλύσει την κατάσταση την οποία παρουσιάσαμε. Γιατί η εφαρμογή, η ερμηνεία και η εισαγωγή της νομοθεσίας αυτής από την ΑΕΝΑ που είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες ελέγχου ε, δεν οδηγεί σε κοινωνική ειρήνη γιατί υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ελλείψεων και παραλήψεων από την πλευρά της ΑΕΝΑ σε σχέση με αυτές τις διατάξεις και έχουμε ένα έγγραφο το οποίο έχει 61 σελίδες που περιλαμβάνουν τις ελλείψεις της εφαρμογής αυτής. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας έχουν οδηγήσει πέραν των νομικών ελλείψεων που έχουν καταγραφεί στις αναφορές μας και έχουν επαληθευτεί από την Eurocontrol αυτά τα οποία καταγγέλουμε, ότι έχουμε έρθει σε μια κατάσταση απόλυτης ανασφάλειας στην εργασία μας που έχει αρνητικό αντίκτυπο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, Ισπανούς ή μη Ισπανούς, που χρησιμοποιούν τις τον Ισπανικό εναέριο χώρο. Ο κύριος Ρουι έχει παρουσιάσει τα στοιχεία, τα οποία είναι συντριπτικά, αλλά αυτά είναι τα στοιχεία της Eurocontrol και όχι τα δικά μου. Μία από τις πολλές νομικές τροποποίησεις που υπέστημεν φέτος έχει να κάνει με την αλλαγή σε σχέση με την μέγιστη, μέγιστο χώρο, ετήσι, μέγιστο χρόνο ετήσιες εργασίας. Με την ε, αλληλουχία των βαρδιών, γιατί η εργασία μας λειτουργεί με εναλλαγή βαρδιών για να μπορεί να υπάρχει υπηρεσία καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Όλα αυτά λοιπόν έχουν τροποποιηθεί από την κυβέρνηση με στόχο την ορθολογικοποίηση του κόστους υπηρεσίας. Και όπως φαίνεται και από τα μέσα ενημέρωσης, και πάλι σας παραπέμπω στο έγγραφο αυτό το οποίο μπορείτε να το αναδυφίσετε όποτε θέλετε, ότι τα μέτρα αυτά δεν είχαν σαν στόχο. Η κυβέρνηση έλεγε ότι όλα αυτά οφείλονται σε κακή διαχείριση. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή επαρκών ελεγκτών για να καλύψουμε τις ανάγκες του εναρίου ελέγχου. Όλες αυτές οι αλλαγές που έχουν να κάνουν με τον χρόνο εργασίας και οι πιέσεις που προέρχονται από την κυρία από την ΑΕΝΑ, όπως είπε ο κύριος Σουηπέρες, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Το προηγούμενο καλοκαίρι ένα σενάριο ελεκτή και είναι πραγματικό αυτό. Το περασμένο καλοκαίρι δουλεύοντα συνέχεια σε Σαββατοκύριακα, νύχτες και τα λοιπά, εργάστηκε κατά, κατά περιτροπή 65 μέρες χωρίς περαιτέρω διακοπές, από μόνο δύο μέρες διακοπές, εργάστηκε 65 μέρες εκτός από δύο μέρες και 29 μέρες χωρίς καμία διακοπή. 63 από τις 65 μέρες λοιπόν και μαζί με τις νύχτες. Χωρίς να υπάρχει λοιπόν καμία μελέτη για τα θέματα ασφάλειας και παραβιάζει αυτό και τον κανονισμό του 93-95. Επίσης είναι γεγονός ότι θεωρεί η ΑΕΝΑ ότι ένας και μόνο ελεγκτής μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του ελέγχου των υπεριπτάμενων αεροσκαφών αλλά και των αεροσκαφών που προσεγγίζουν ένα κέντρο ελέγχου στην περιοχή των Κανάριας και άλλων. Αυτό είναι κάτι ε, οδήγησε στο ατύχημα του 2002 πάνω από την ε, Μπόντενζέ, από τη λίμνη της Κωνσταντζας, στο οποίο σκοτώθηκαν 71 άτομα. Επίσης, προβλέπεται ότι μπορεί ένας ελεκτής να κληθεί να εργάζεται τις ημέρες ε, ανάπαυσής του. Και αυτοί οι οποίοι αρνούνται έχουν να αντιμετωπίσουν κυρώσει διοικητικές και οικονομικές πρόστιμα τα οποία φτάνουν σε χιλιάδες ευρώ. Όλο αυτό παραβιάζει το βασικό δικαίωμα κάθε εργαζομένου να εργάζεται σε συνθήκες οι οποίες είναι ισοδίκες και σας λέω και πάλι ότι όλα αυτά μειώνουν την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της ενέργειας ασφάλειας, πιέζουν ιδιαίτερα την υγεία τους σε σωματικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο λόγω της υψηλής πίεσης και αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα την ασφάλεια των, ε, της ενέργειας κυκλοφορίας. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση και η ΑΕΝΑ προσπαθούν να τα ε, απορρίψουν. Είναι σαφή τα στοιχεία αυτά, υπάρχουν αυτές οι επιπτώσεις στην ενέργεια ασφάλεια τα οποία αναφέραμε και υπάρχει και το γεγονός ότι κατά 350% έχουν αυξηθεί καθυστερήσει στον ενάριο έλεγχο σε σχέση με το 2008 που ήταν το έτος στο οποίο υπήρχαν οι περισσότερες ε, πτήσεις. Σε ένα χρόνο λοιπόν που έχει μικρότερη εναέρια κίνηση έχουμε πολύ περισσότερες ε, καθυστερήσεις από το 2008 που ήταν το έτος με τις περισσότερες κινήσεις. Και έχουν αυτή τη στιγμή οι οι πτήσεις στην Ισπανία να είναι στην πρωτοπορία των πιο ανασφαλών πτήσεων και των πτήσεων που έχουν ακόμα από πιο μεγάλες καθυστερήσεις. Ο υπέτειος πρέπει να ζητηθεί στις τάξεις της Ισπανικής κυβέρνησης. Όπως έλεγε και ο συνάδελφός μου, τι λύση μπορούμε να δώσουμε στα θέματα αυτά. Εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ενάρεια συμφόρηση, επομένως ο μεγαλύτερος κίνδυνος ε, ατυχημάτων, έχουμε έχει ζητήσει η ΑΕΝΑ να υπάρξει μικρότερος αριθμός ελεκτό και έχει ζητήσει η απόσταση μεταξύ των αεροσκαφών στους αεροδιαδρόμους. Σας ζητούμε λοιπόν να λάβετε όλα τα μέτρα τα οποία περνούν από το χέρι σας για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Είναι 200 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που πετούν πάνω από την Ισπανία κάθε χρόνο. Δεν είναι μοναχανικό πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου. Επομένως θα πρέπει να δράσετε με ταχύτητα και με αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Μάιερ. Πριν σας δώσω, πριν δώσω το λόγο στους βουλευτές για τη συνέχιση του διαλόγου. Δίνω το λόγο στον κύριο Δημητρίου από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει πραγματικά τις προσφυγές των αναφερόντων όχι μόνο στα πλαίσια της αναφοράς που υπευλήθη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στα πλαίσια επιστολών και διαμαρτυριών που έφτασαν κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν επίσης να σας πω ότι στις 27 Ιουλίου 2009 εστάλει και μία επιστολή. Κατόπιν το Νοέμβριο του 2010 ο κύριος Σιλ ο ίδιος έστειλε μια επιστολή που παρουσιάζει όλα αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο αυτά που περιλαμβάνονται εδώ σε αυτήν την αναφορά, αλλά και όλες τις υπόλοιπες ε, διαμαρτυρίες. Γι' αυτό και θα ήθελα να πω ότι στην Επιτροπή εστάλει μετά την επιστολή αυτή του Νοεμβρίου. Υπάρχει ένα διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, μια προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για τους ε, αναφέροντες, για σχόλια. Δεν λάβαμε λοιπόν σχόλια, γι' αυτό και έκλεισε το θέμα στην Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά το διαδικαστικό κομμάτι, Επί της ουσίας όμως που μας παρουσίασε ο αναφέρον, άκουσα πολύ προσεκτικά τα διαφθόρα σημεία που αναπτύξατε και που μας παρουσιάσατε εδώ και ήθελα να πω ότι δεν θα επαναλάβω τα ίδια και τα ίδια. Ξέρετε ότι η Επιτροπή έχει κάνει δύο ε, δηλώσεις, δύο ανακοινώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτές τις έχετε εξάλλου μεταβιβάσει και στους αναφέροντες. Και έχουμε απαντήσει εις μάθος τα διάφορα σημεία που υπογραμμίζουν οι υπογράφοντες την αναφορά. Θα κάνω κάποια γενικά σχόλια καταρχήν. Όντως, τα θέματα αυτά αναφέρονται σε πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα, τα οποία είναι αντιφατικά τα οποία έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση. Παραδείγματο χάρη υπάρχει η κατάσταση στην ενέργεια κυκλοφορία. Δεύτερον, οι συνθήκες εργασίας στο χώρο της ενέργειας κυκλοφορίας. Και αυτό αφορά όχι μόνο την Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, αλλά και τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αυτές οι απαντήσεις έχουν ήδη υποβληθεί από την Επιτροπή στους αναφέροντες. Θέλω επίσης να πω ότι τα θέματα που θίξατε αφορούν και κάποιες γραπτές ερωτήσεις. Παραδείγματο χάρη, το θέμα της απεργίας που έλαβε χώρα στην Ισπανία πριν από λίγο καιρό Αυτό αναφέρεται και σε κάποιες από τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως όλοι ξέρετε, που έχουν μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως όλοι ξέρετε εξάλλου. Τώρα, το δικαίωμα του συνέρχεστε το δικαίωμα των ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων και βεβαίως οι συνθήκες και βεβαίως η συνθήκη της Λισαβόνας έχουν δημιουργήσει σήμερα μια νομικά δεσμευτική κατάσταση. η συνθήκη της Λισαβόνας έχει ενσωματώσει, όπως ξέρετε, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό βεβαίω δεν σημαίνει ότι είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα αυτό. Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ένα από τα άρθρα του αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν νομοθετεί πρέπει να λαμβάνει υπόψη το αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ίδια ώρα αφορά τα κράτη-μέλη μόνο και εφόσον τα κράτη-μέλη μεταφέρουν και εφαρμόζουν κοινοτικό δίκαιο. Εξού και δεν καλύπτονται οι αναφέροντες από κοινοτικό δίκαιο. Αναφέρατε μία σειρά οδηγιών. τις οποίες αναφέρατε ως ε, εφαρμόσιμες, ως αρμόδιες, ως οδηγίες που μπορείτε να επικαλεστείτε για αυτές τις υποθέσεις. Δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες των απαντήσεών μας, αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες από αυτές τις οδηγίες. Είπατε ότι υπάρχουν νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν φαίνονται να εφαρμόζονται εδώ. 2002 κάθετος 14 όσον αφορά την συμμετοχή των εργαζομένων σε μια απόφαση που δεν αφορούν όμως τις συλλογικές συμβάσεις, δεν μπορούν να εφαρμοστούν εδώ. Οδηγία 2000 κάθετος 78 για την έλλειψη διακρίσεων, αποφυγή διακρίσεων και εδώ δεν αναφέρεται το θέμα αυτό στις διακρίσεις, αλλά έχετε δίκιο και υπάρχουν κάποια άλλα θέματα που καλύπτονται από άλλες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραδείγμα χάρη το θέμα τη υγιεινής και ασφάλειας στον τόπο εργασία. Τουλάχιστον εδώ έχουμε ένα οπλοστάσιο νομικών ε, εργαλείων και μέσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν το θέμα αυτό. Η 2003 κάθετος 33 και η γενική, η οδηγία πλαίσιο για την υγιεινή και την ασφάλεια. Όπως σας είπα, δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες αυτών των νομικών κειμένων όσον αφορά την συμβατότητα αυτών των κειμένων με τα όσα επικαλείστε. Όσον αφορά το χρόνο εργασίας, παραδείγματος χάρη, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει εδώ θέμα συμμόρφωσης και όσον αφορά το θέμα αυτό θεωρούμε ότι αρμόδιες είναι οι εθνικές αρχές για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Αυτό που στην παρουσίασή σας είναι διαφορετικό σήμερα είναι ο νέος νόμος του Μαρτίου. Εμείς πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε λάβει γνώση αυτού του νέου νόμου Άρα δεν μπορούμε να τον έχουμε εξετάσει και δεν μπορούμε να πούμε εάν είναι συμβατό το κείμενο του νόμου αυτού με τον κοινοτικό νόμο. Πρέπει να σας πω ότι αναφέρατε ένα κείμενο 60 σελίδων Δεν γνωρίζω όμως ε, το κείμενο του νόμου αυτού. Δεύτερον, σημείωσα το παράδειγμα που αναφέρατε, τον συνάδελφό σας, ο οποίος εργαζόταν 65 μέρες χωρίς καμία άδεια. Αν σημειώσα καλά, είπατε ότι εργαζόταν συνέχεια επί 29 ημέρες, χωρίς καμία απολύτως άδεια. Εδώ δεν τίθεται μόνο θέμα εφαρμογής του κοινοτικού νόμου. Εδώ είναι καθαρά θέμα βεβαίως ε, των εθνικών αρχών. Θα έπρεπε ο επιθεωρητής εργασίας, ο Ισπανός, να είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό, γιατί πρόκειται για μη εφαρμογή ή κακή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Και βεβαίως βάσει συγκεκριμένων γεγονότων μπορούμε να ε, πάρουμε θέση εδώ. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι τα θέματα της ασφάλειας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι επίσης θέμα συζητήσεων στην Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου. Οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στην συζήτηση αυτή, αλλά και η DG Move, Γενική Διεύθυνση Κυκλοφορία, έχει σημειώσει τα διάφορα σχόλια. Εξάλλου αναφέρθηκα και προηγουμένως στις απαντήσεις που πρέπει να έχετε λάβει από μέρους της Επιτροπής που συμπεριλαμβάνουν αυτά τα σχόλια. Κυρίως το κατά πόσο υπάρχει ή δεν υπάρχει συμμόρφωση ή συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, ιδιαίτερα η DG Move, συμπεραίνουν ότι είναι θέμα των εθνικών αρχών να εξετάσουν όλα αυτά τα θέματα που προκύπτουν σε σχέση με την συμβατότητα και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο κάλυψα σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα σημεία που μας παρουσιάσατε σήμερα. Αλλά βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας εάν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τουργκάης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ καλά γνωστό στη χώρα μας, στην Ισπανία. Όταν ακούσαμε τους ε, αναφερόμενους να μας εξηγούν την κατάσταση, και ότι ήδη η Επιτροπή τους, ε, τους απήντησε ότι αυτό είναι ένα θέμα εθνικού χαρακτήρα και ότι αυτό πρέπει να επιληθεί μέσα στο ισπανικό πλαίσιο και το Ισπανικό Κοινοβούλιο και το, τα Ισπανικά δικαστήρια πρέπει να δώσουν μια λύση. Όταν είδα αυτή την ε, αναφορά ήδη πριν από κάποιο χρόνο, πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, εγώ είχα πει ότι πρέπει αυτή η ασφάλεια να δεν επιχειρηματολογούσε επί της ε, βάσης της ε, εργατοργασίακων εργασιακών συνθηκών αλλά και επί τη βάση της ενέργειας ασφάλειας. Είναι πραγματικά ανησυχητικά τα στοιχεία αυτά τα οποία έχετε αναφέρει γιατί καταδεικνύουν σύμφωνα με τη δική σας επαγγελματική άποψη ότι υπάρχει μια σοβαρή ασφάλεια, έλλειψη ασφάλειας στους ισπανικούς εθέρες και αυτό σημαίνει και στους ευρωπαϊκούς εθέρες. Ενώπιον λοιπόν αυτών των θεμάτων που είναι πάρα πολύ σημαντικές καταγγελίες και σίγουρα όπως είπατε εσείς υποστηρίζονται και από έγγραφο της ε, Eurocontrol θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα στην Κομισιόν αν, για το αν η Κομισιόν έχει τα στοιχεία αυτά τα οποία αναφέρθηκαν οι αναφερόμενοι για την έλλειψη ενέργειας ασφάλειας που έχουν ένα ανησυχητικό χαρακτήρα ή θα έπρεπε να μας ανησυχούν όλους μας, όχι μονάχα για τον Ισπανικό ενάριο χώρο, αλλά και τον Ευρωπαϊκό χώρο. Καταρχήν λοιπόν το πρώτο ερώτημά μου είναι αν είναι εν γνώση η Κομισιόν αυτής της έλλειψης ασφάλειας, αν γνωρίζει όλα αυτά τα στοιχεία. Και το τρίτο σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω, τι θα πράξει σχετικά η Κομισιόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας που χρησιμοποιούμε, την, ε, χρησιμοποιούμε αεροπλάνα σε καθημερινό επίπεδο. Τι θα κάνει λοιπόν η Κομισιόν για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ Έχω ακούσει ένα από τους αναφερόμενους να λέει ότι ζητάει από την Επιτροπή Αναφορών να λάβουμε όλα τα μέτρα τα οποία περνάνε από τα χέρια μας. Και τώρα βρισκόμαστε και πάλι σε μια κατάσταση όπου δεν κατανοούν οι αναφερόμενοι τι ρόλο παίζει η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν είμαστε ένα δικαστήριο. Δεν είμαστε ένας φορέας στον οποίο έρχεται κάποιος και δίνει λύση σε κάτι. Είναι ένας φορέας με τεράστια ε, υπομονή. Αυτό είναι γενικό. Είναι γενική κρίση. Έχουμε, έχουμε μεγάλη υπομονή και είμαστε πάντα έτοιμοι να ακούσουμε τους αναφερόμενους. Αλλά στο τέλος λέτε εμείς διεκδικούμε το α, το β, το γ. Δεν μπορεί να σας δώσει καμία απάντηση στις διεκδικήσεις σας. Η Επιτροπή Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι ένας φορέας ο οποίος θα σας πει συμφωνώ διαφωνώ με αυτά που λέτε. Δεν έχει καμία ικανότητα, δεν έχει καμία ευθύνη εξάλλου για να δώσει απάντηση στον κατάλογο των διεκδικήσεών σα. Κάποιες είναι συνδικαλιστικού χαρακτήρα, κάποιες δεν είναι λοιπά. Δεν θα μπω λοιπόν σε λεπτομέρεια στις ε, δηλώσεις και τις καταγγελίες σας που πιστεύω ότι είναι μεροληπτικές στην καλύτερη περίπτωση. Αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν, αυτά που δεν δημοσιεύτηκαν, το πώς, σε ποιες συνθήκες δημοσιεύτηκαν, οι αμοιβέ των ε, ελεγκτών που συγκρίθηκαν με τις, ε, τις αμοιβέ άλλων ελεκτών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η κατάσταση ορισμένων συναδέλφων που είχε να εργάζεται υπερορίες και όταν ήταν οι υπερορίες που πληρωνόντουσαν δεν ένιωθε στρες αλλά όταν γινόντουσαν οι υπερορίες Κανονικέ ώρε ένιωθε ένα πολύ μεγάλο στρε και μεγάλη πίεση. Δεν θα πω τώρα σε αυτά τα επιχειρήματα. Γιατί εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά θέματα. Και το είπε πολύ σωστά η Κομισιόν. Από τη μία πλευρά μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι θέμα εργασιακό και από την άλλη πλευρά για ένα θέμα το οποίο είναι θέμα ασφαλεια Και επιμένω και πάλι για να το καταλάβουν και οι αναφερόμενοι. Αν θέλουν να επιτύχουν κάποια λύση στο πρόβλημά του. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία είναι θεμητό να τους απασχολούν. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών ότι δεν υπάρχει παραβίαση κοινοτικών κανόνων, αυτή η αναφορά θα πρέπει αυτομάτως να εξαλειφθεί από την ημέρησια διάταξή μας. Γιατί ο ρόλος μας είναι να ακούσουμε και να ακούσει η Κομισιόν φυσικά, όπως είπε ο κ. Σιτουργκάης, για το αν θεωρεί η Κομισιόν ότι υπάρχει παραβίαση ή όχι του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου. Δεν βρισκόμαστε στην Πουέρτα Δελσό, δεν βρισκόμαστε στον χώρο που ο βασιλιάς απονέμει χάρη ή δέχεται τις αναφορές των πολιτών. Είμαστε η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν λοιπόν δύο περιοχές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η μία είναι το, τα εργασιακά θέματα και φαίνεται ότι μετά από πάρα πολύ χρόνο διαπραγματεύσεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας όλα αυτά που έγιναν έγιναν με ένα τρόπο ο οποίος ε, έγινε σύμμορφα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλήξαμε σε μια συμφωνία μεταξύ των ε, συνδικάτων και των εργοδοτών και η οποία επικυρώθηκε από ένα 85% των εργαζομένων στον τομέα αυτό. όλοι μας που έχουμε σταθεί συνδικαλιστές στο παρελθόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί πάντα, γιατί το αποτέλεσμα μιας διαιτητικής λύσης δεν είναι πάντα κάτι το οποίο μας ικανοποιεί. Μας φέρνει πολλές φορές ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι αυτό το οποίο επιζητούσαμε αλλά έγινε δεκτή αυτή η λύση από την πλειοψηφία των εργαζομένων. Για μένα λοιπόν έχει κλείσει το θέμα αυτό. Αυτό το οποίο με απασχολεί όμως πάρα πολύ είναι αυτά τα οποία ελέγχθηκαν για την εναέρια ασφάλεια. Και εγώ επιτρέπω στον εαυτό μου να πω ότι το ίδιο αυτό έγγραφο το οποίο αναφέρεται της ε, Eurocontrol δεν είναι αυτό το οποίο αναφέρεται από ορισμένου κύκλους της άκρας δεξιάς. Το έγγραφο της Eurocontrol λέει περίπου τέσσερις φορές για τα κύρια σημεία ότι τα στοιχεία αυτά τα οποία δίνονται δεν είναι αξιόπιστα. Και λέει επίσης υπάρχει έλλειψη συνεκτικότητος στην, στις εκθέσεις και στην ε, αναφορά των επεισοδίων και δεν επιτρέπει στη Eurocontrol να εντοπίσει και να ε, διαπιστώσει τάσεις για τα θέματα αυτά. Στο τρίτο σημείο λέει επίσης ο αριθμός των παραβιάσεων ελάχιστης απόστασης μειώθηκε κατά 20% το 2008 επί τη βάση επιβεβαιωμένων στοιχείων και μειώθηκε κατά άλλα 44% το 2009 επί τη βάση προσωρινών στοιχείων. Αλλά η έλλειψη συνέπειας σε σχέση με τις αναφορές για τα προβλήματα αυτά παραβίασης ελάχιστης απόστασης δεν, υπάρχει, δεν δίνει δυνατότητα στη Eurocontrol να έχει μια σαφή αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά. Τέταρτο σημείο. Ο αριθμός των εισβολών στον, στους αεροδρόμους μειώθηκε το 2008 και κατά 7% το 2009. Ο αριθμός των ε, εισβολών σε αεροδρόμους που δεν εξετάστηκαν το 2009 παραμένει πάρα πολύ υψηλός για να μπορείς κανείς να παρακολουθεί την πορεία των στοιχείων. Αυτά λέει το Eurocontrol. Δεν είναι ένα έγγραφο το οποίο έχω γράψει εγώ. Και τούτου λεχθέντος Θέλω να σας πω ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, νομίζω ότι ορισμένε από τις δηλώσει που έχουν γίνει εδώ, και όχι μόνο ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών που έχει αυτές τις ευθύνε που έχει, αλλά και ενώπιον της Ευρωπαϊκής ε, των Μέσων Ενημέρωσης, είναι κάπως κινδυνολογικές, μη εμπεριστατωμένες και ανεύθυνες. Και δυνητικά πάρα πολύ επικίνδυνε για τα συμφέροντα της χώρας μου. Θέλω λοιπόν να το κάνω απόλυτα σαφέ για όλους τους συναδέλφους. Γιατί πάνω απ' όλα εμείς ως Ευρωβουλευτές είμαστε από του κύριους χρήστες των εναερίων μέσων μεταφοράς. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι είναι κινδυνολογικές, είναι βεβαιασμένε, είναι ανεύθυνε και δυνητικά πάρα πολύ αρνητικές για τα συμφέροντα τη χώρας μου. Θέλω να τονίσω λοιπόν, αυτό είναι ο χαρακτήρα των δηλώσεων αυτών, εγώ τι ε, δέχομαι, αλλά εποφελία απογραφής και με πάρα πολύ μεγάλε επιφυλάξει και αναμένω την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βασίζομαι σε αυτά τα οποία μας είπε σε σχέση με την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, την παραβίαση. Αυτά με κάθε σεβασμό για αυτούς οι οποίοι ήρθαν να μας εκφράσουν τις απόψεις τους. Δεν ξέρω αν ήρθαν με λανθασμένη εντύπωση ότι εδώ θα, θα λυθούν τα προβλήματά τους ή με την ε, πρόθεση να κάνουν απλώς δώρο και να βγουν τα θέματα αυτά στα, μέσα ενημέρωσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα τρει παρεμβάσει και πρέπει κάποια στιγμή και να τελειώσουμε, γιατί έχουμε και την ε, συνάντηση των συντονιστών. Ο κύριο Μέγερ, παρακαλώ να είστε πιο σύντομο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω αυτού οι οποίοι παρουσίασαν τι αναφορέ αυτέ. Υπάρχει ένα τμήμα τη αναφορά που είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε, που έχει να κάνει με την εργασιακή σύγκρουση που έλαβε χώρα στην Ισπανία. Η Σκέρδα Ουνίδα, η πολιτική ε, παράταξη που εγώ υποστηρίζω κατηγορήθηκε για μια στρατικοποίηση αυτής της ε, σύγκρουσης. Εμείς δεν ήμασταν αντίον της ε, συμπερίληψης των ε, ελεγκτών στην ΑΕΝΑ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να θεωρείς κανείς ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν στον εργασιακό χώρο είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Υπάρχει λοιπόν ένα τμήμα αυτών των πληροφοριών που Κύριε Μαρτίνες όμως θα συμφωνήσετε ότι δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι αυτή την πληροφόρηση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη διαλεύκανση για τα θέματα αυτά. Γιατί εσείς με αυτά που είπατε θέτετε εν την εναέρια ασφάλεια στον Ισπανικό εναέριο χώρο και στον Ευρωπαϊκό εναέριο στους ε, ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες. Γι' αυτό θα πρότεινα σε σχέση με το θέμα αυτό να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αναμένοντας να έχουμε μια επιβεβαίωση ή μια διάψευση αυτών των στοιχείων. Η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί χωρίς κατά αντιμολία διαδικασία, χωρίς να έχει έγκυρες πληροφορίες, δεν μπορεί να κλείσει αυτή την αναφορά. Αν μου επιτρέπει λοιπόν και η κυρία Άουκεν, ζητώ επισήμως η Επιτροπή μας να κρατήσει ανοιχτή αυτή την αναφορά για το τμήμα της Ενάρειας ασφάλειας και να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση η οποία θα παρουσιάσει και τις δύο απόψεις για τα θέματα της Ενάρειας ασφάλειας των Ισπανικούς εθέρες. Κύριε Πρόεδρε, σαν μέλος της Επιτροπής Αναφορών, πιστεύω ότι έχουμε περιορισμένους τρόπους να αντιδράσουμε περιορισμένα μέσα. Σαν μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης, φυσικά και με απασχολεί πολύ το θέμα αυτό των συνθήκων εργασίας των ε, ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας στην Ισπανία. Σαν πιλότος ε, εγώ ίδιος χαίρομαι γιατί συνειδητοποιώ ότι όταν ε, περνάω μέσα από τον εναέριο χώρο της Ισπανίας κινδυνεύει η ζωή μου και από εδώ και πέρα θα προσπαθώ να αποφεύγω αυτόν τον εναέριο χώρο ακούγοντας τον κύριο Μάγερ ο οποίος ζητάει να παραμείνει το θέμα αυτό ανοιχτό θα συμφωνήσω μαζί του και πιστεύω ότι όπως προτείνει η Επιτροπή ίσως πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε βασιζόμενοι στα στοιχεία Eurostat ο κύριος Μαρτίνης λέει κάποια πράγματα οι αναφέροντες ε, έχουν διαφορετικά στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει με θέματα υγείας των ε, ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας στην Ισπανία αλλά και ασφάλειας όσον αφορά την ενέργεια κυκλοφορία στην Ευρώπη, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό που υποτίθεται ότι αυξάνει την ασφάλεια με ενιαία στοιχεία. Πολύ σύντομα, γιατί έχουμε περάσει τρία τέταρτα να το συζητάμε αυτό και το βρίσκω παράλογο. Γιατί είναι αμφίβολο αν η αναφορά αυτή ευσταθεί και είναι παραδεκτή για την Επιτροπή μας. Όπως έχει διατυπωθεί, είναι εθνικό το θέμα, αλλά θέτει και ζητήματα ασφάλειας. Ας σταματήσουμε εδώ την συζήτηση και ας αφήσουμε το θέμα ανοιχτό, αλλά είναι πραγματικά παράλογο να έχουμε περάσει τόσο πολύ χρόνο για μια τέτοια αναφορά. Και κάτι που έχει ξανασυμβεί η δυσκολία μας είναι ότι οι αναφερόμενοι, οι πολίτες, δεν καταλαβαίνουν τελικά ποιε ακριβώ είναι οι αρμοδιότητέ μα και δεν μπορούν να τι διακρίνουν από τι εθνικέ. Εδώ σταματάω. Σταματάω. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με όλη αυτή την κουβέντα. Ευχαριστούμε κυρία Οκέν. Ένα λεπτό για την κάθε απάντηση. Ένα και ένα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, ακόμα και στα όρια του αδυνάτου. Για τον κύριο Μαρτίνες θέλω να πω το εξής είπε ότι εμείς θεωρούμε ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι ένας χώρος όπου πηγαίνουν οι αγανακτισμένοι και ζητούν τα δικαιώματά τους. Όχι. Εμείς βασιζόμαστε στο βασικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κάτι το οποίο είναι απαράγραπτο δικαίωμα του κάθε πολίτη η Επιτροπή σας είναι μια Επιτροπή η οποία μπορεί να κάνει έρευνες, μπορεί να ζητήσει εξοδικαστικές λύσεις. Αυτά λέει η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια Επιτροπή που μπορεί να ερευνήσει και μπορεί να βρει λύσεις ε, εξοδικαστικού χαρακτήρα για, τα, για τις καταγγελίες μας. Μπορεί να οργανώσει επισκέψεις έρευνες και να πληροφορήσει την Ολομέλεια, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρξει εγκύτητα προς τους πολίτες και να ενισχυθεί η δημοκρατική νομοποιηση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι η Επιτροπή ε, Αναφορών είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να δώσει κάποιες ε, λύσεις και όχι ένας χώρος όπου απλώς διατυπώνουμε τα αιτήματά μας. 30 δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, πάρα πολύ συγκεκριμένο. Το εξής η απάντηση που πήραμε από την Κομισιόν μέσα, μέσω του κυρίου Δημητρίου οδήγησε και σε μία προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπαν λοιπόν και οι συνάδελφοι, εμείς ε, πληροφορήσαμε τον κύριο Σίμ Κάλλας και τα, τα μέλη του γραφείου της κυρίας Ρέντινγκ τονίζοντας ότι υπάρχει ένα σημαντικό θέμα για την ενέργεια ασφάλιση. Ο κύριος Μακμίλαν επίσης από το Eurocontrol το γνωρίζει το θέμα αυτό. Ο κύριος Στόιον μας ζήτησε να δώσουμε αντίγραφο των ε, δηλώσεων των 1.300 ε, ενέργειων ελεγκτών που θεωρούν ότι εργάζονται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Ναι, για το σημείο της ασφάλειας. Έχει έρθει στη γνώση όλων των συναδέλφων και θα το εμβαθύνουμε. Σας παρακαλώ. Δεν είναι η Υπηρεσία Κοινωνικών Υποθέσεων, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων που πρέπει να απαντήσει σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Σε 30 δευτερόλεπτα απαντώ στα στοιχεία που έδωσε ο κ. Μαρτίνες. Όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν μια μείωση των επεισοδίων είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρώπη μειώνονται τα επεισόδια, στην Ισπανία αυξάνονται. Είναι η ίδια ακριβώς έκθεση που εγώ ανέφερα και μου λέτε ότι είναι χωρίς βάση όλα αυτά που σας λέω. 47 επεισόδια τύπου Α και 90 τύπου Β. Είναι μια ανακοίνωση της ΑΕΝΑ. Βρίσκεται μέσα στην έκθεση performance report του Eurocontrol που βγήκε πριν από μια εβδομάδα. Δεν φαντάζομαι πράγματα, δεν τα επινοώ εγώ. Είναι πραγματικότητα. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι επειδή λέτε ότι επειδή μας έχουν καταπατήσει τα εργασιακά δικαιώματα, ότι εμείς τώρα θέτουμε την ασφάλεια σε κίνδυνο επίτηδες. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Θέλω επίσης να απαντήσω και στην Κομισιόν. Οι εθνικές αρχές έχουν χιλιάδες καταγγελίες για την κατάσταση αυτή και περιμένουμε ακόμα να πάρουμε απάντηση από αυτές. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστούμε. Η, αυτή, η αναφορά αυτή παραμένει εντύπωση. Θα ζητήσουμε λοιπόν περαιτέρω μελέτη σε σχέση με την διάσταση της ασφάλειας. Ίσως το συζητήσουμε και στη συνεδρίες των συντονιστών ποια είναι η καταλληλότερη οδό. Κλείνουμε την συνεδρίαση αυτή. Παρακαλώ να βγουν οι ε, προσκεκλημένοι για να ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών.